Συνάδελφοι, είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Είμαστε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, πρώτο σημείο, παρουσίασε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση ε, στην οποία βρίσκονται τα μέτρα διασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Χάλιβα. Θα θυμάστε ότι μετά από τα μέτρα που, επέβαλε η, που επέβαλαν οι ΙΠΑ στο αλουμίνιο και το χάλιβα, ε, δημιουργήσαμε κι εμείς ένα σύστημα διασφάλισης, μέτρων διασφάλισης, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τη δική μας τη βιομηχανία χάλιβα. Από τις συνέπειες των μέτρων των ΙΠΑ. Η Κομισιόν θα υποβάλει τη γνωμοδότησή της το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου και θα πρέπει να συζητήσουμε, να δούμε αν αυτά τα μέτρα διασφάλισης είναι αποτελεσματικά και αν θα πρέπει να βελτιωθούν. Αυτό θα είναι το πλαίσιο της συζήτησης σήμερα, οπότε δίνω το λόγο στην Κομισιόν να μας παρουσιάσει τα δεδομένα και το πώς έχει η κατάσταση. Ο Λεοπόλντο, ο φίλος μας, θα μας κάνει την παρουσίαση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Όντως, η Κομισιόν υιοθέτησε αυτά τα μέτρα διασφάλισης σε 26 κατηγορίες προϊόντων χάλιβα στις 2 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους τα μέτρα, όπως ξέρετε, όπως είπατε πολύ σωστά, υιοθετήθηκαν μετά από κάποιες πολύ ενσυχητικέ ε, ε, εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά χάλιβα και τη θέση των, που έλαβαν οι ΙΠΑ στον τομέα 232 για τον ε, χάλιβα. Και βεβαίω υπήρξαν και κάποια περιοριστικά μέτρα επί του Χάλιβα που είχαν επιβληθεί από άλλου εμπορικού μα εταίρου. Βεβαίω, οι νομικέ απαιτήσει για την επιβολή τέτοιου είδου μέτρων τηρούνται. Κυρίω ε, διαπίστωσε η Κομισιόν ότι από, την περίοδο από το 2013 έω το 2017 υπήρξε απόλυτη αύξηση εισαγωγών ε, προϊόντων χάλιβα, πολύ μεγάλη μάλιστα αύξηση σε μερικές περιπτώσεις και το πιο σημαντικό είναι ότι η Κομισιόν διαπίστωσε ότι ως αποτέλεσμα αυτών των δραστικών αυξήσεων η ευρωπαϊκή βιομηχανία μπορεί να ε, απειλείται με σημαντικές ζημίες. Οπότε, ε, και ε, τονίζω εδώ τον όρο απειλείται, διότι ήταν σημαντικό να δράσουμε πριν βεβαίως πληγεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ο βασικός στόχος των μέτρων διασφάλισης είναι να αποφευχθεί ε, διαφοροποίηση του εμπορίου μετά από το κλείσιμο της ε, αμερικανικής αγοράς αλλά και άλλων ταυτόχρονα προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε τις παραδοσιακές εμπορικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επαρκή ασφάλεια της τροφοδοσίας. Είναι σημαντικό επίσης να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτάρκης σε χάλιβα, πρέπει να εισάγει και επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη ότι και οι 26 κατηγορίες αυτών των προϊόντων που υπόκεινται στα μέτρα είναι επίσης ε, υλικά και, προς και κατάντι στην βιομηχανία, έτσι όπως αυτή ε, λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ήταν ιδιαίτερο σημαντικός για μας να έχουμε μια ισόρροπη προσέγγιση και να φροντίσουμε να ε, καλύψουμε όλα τα κενά. Έχουμε 150 μέρη που συμμετέχουν στην όλη έρευνα, 93 ακροάσεις έλαβαν χώρα και στο τέλος αυτής της αρκετά περίπλοκης διαδικασίας αποφασίσαμε να επιβάλλουμε μέτρα με τη μορφή ε, δεσμολογικών ποσοστώσεων, πάνω από την οποία ε, επιβάλλεται ένα 25% τέλος. Επίσης αποφασίσαμε να εξεύρουμε έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε, χωρίς όμως να διακυβεύσουμε την ασφάλεια της τροφοδοσίας. Και επίσης θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι οι παραδοσιακές εμπορικές ροές θα ε, γίνουν σεβαστές χωρίς βεβαίως να υπάρχει αποθεματοποίηση ή ε, κερδοσκοπία. Και γι' αυτό ε, αποφασίσαμε να βάλουμε δοσμολογικές ποσοστώσει ανά χώρα για τους ιστορικούς παρόχου τη αγορά, αυτούς δηλαδή που καλύπτουν 25% της αγορά και κάποιε εναπομείνασε ποσοστώσει για του υπόλοιπου. Αυτέ οι ποσοστώσεις θα είναι διαθέσιμες για όλους από το τέταρτο τρίμηνο κάθε περίοδου. Τα προσωρινά μέτρα μπήκανε τον, επιβλήθησαν τον Ιούλιο. Άρα το τέταρτο τρίμηνο ξεκινάει 1η Απριλίου. Χτες λοιπόν ξεκίνησε το, το τέταρτο τρίμηνο της ε, ε, συνολικής αυτής ε, ποσόστοσης. Ελέγχουμε τη χρήση των ε, δοσμολογικών ποσοστώσεων καθημερινά. Η, ο τρόπος ε, ελέγχου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ταξούντ και μέχρι στιγμής θεωρούμε ότι η χρήση των ποσοστώσεων δεν παρουσιάζει προβλήματα για την ε, ε, πλειοψηφία των ποσοστώσεων. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι οι ποσοστώσεις δεν χρησιμοποιούνται πλήρως πολλές φορές ε, παρασάγκας απέχουν από το να χρησιμοποιηθούν πλήρως, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, τις οποίες ξέραμε ότι θα είναι προβληματικές βέβαια, και βλέπουμε ότι οι ποσοστώσεις έχουν εξαντληθεί, έχουν φτάσει στο 100%. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν οι εξαγωγοί, οι εξαγωγοί χώρες θέλουν να συνεχίσουν να εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το, 25%, ε, το τέλος αυτό του 25% θα πρέπει να καταβληθεί. Επίσης διαπιστώσαμε ότι ο βασικός μας πάροχος χρησιμοποιεί πλήρω τις ε, ε, προστάσεις και αυτό είναι η Τουρκία. Είναι μια χώρα που μας ε, παρέχει χάλιβα και είναι και μια χώρα που εξάγει πολύ ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρε, όπως είπατε σωστά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε περιοδικώς να αναθεωρεί αυτά τα μέτρα και θεωρούμε ότι η αγορά του Χάλιβα είναι μια πολύ δυναμική αγορά και το να καθορίσουμε για τρία χρόνια συγκεκριμένα μέτρα θα ήταν πολύ μακρά περίοδος. Οπότε αποφασίσαμε ότι θα μελετούμε, θα ελέγχουμε τα μέτρα αυτά σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Η πρώτη αναθεώρηση προβλέπεται να γίνει την 1η Ιουλίου το αργότερο. Αλλά προς το παρόν συζητούμε και εντός των υπηρεσιών της Κομισιόν το κατά πόσο είναι δυνατόν να αρχίσει νωρίτερα η αναθεώρηση, πριν την 1η Ο στόχος της αναθεώρησης αυτής δεν θα είναι να αμφισβητήσουμε τις, ε, ε, τα μέτρα διασφάλισης. Ο στόχος είναι αν, να δούμε αν χρειάζεται προσαρμογή των δασμολογικών ποσοστώσεων. Ας πούμε, επειδή παρατηρήθηκε ότι οι δασμολογικές ποσοστώσει θα πρέπει να, γίνουν, να καταναμηθούν με διαφορετικό τρόπο ή θα πρέπει να τύχουν διαφορετική διαχείριση. Το ουσιώδες εδώ για την επιβολή των οριστικών μέτρων είναι το συμφέρον της Ένωσης. Τι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να κάνει, πρέπει να αλλάξουμε κάτι ή όχι. Ω προ αυτό λοιπόν υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά και πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Το πρώτο, όπω είπα, είναι ότι έχουμε κάποιε δασμολογικέ ποσοστώσει που έχουν εξαντληθεί πλήρω και ήδη έχουμε αντιπροσωπείε από αρκετού εισαγωγεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παραπονούνται για το ότι δεν μπορούν πλέον να ε, παράξουν τα υλικά αυτά και επίση βλέπουμε ότι και κάποιε αναπτυσσόμενε χώρε, όπω η Ινδονησία έχουν αρχίσει να ε, εξάγουν σε μεγάλους όγκους συγκεκριμένα προϊόντα. Όπως ξέρετε, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, οι αναπτυσσόμενες χώρες που αποτελούν κάτω από το 3% των εισαγωγών θα πρέπει να, να εξαιρούνται από, τις... από τα μέτρα διασφάλισης. Όταν κάναμε εμείς τη δική μας έρευνα, χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα που υπήρχαν τότε, δηλαδή τα δεδομένα για το TLD από, το 2000, από τον Ιούνιο του 2018 και η Ινδονησία επί τη βάση εκείνων των δεδομένων δεν περνούσε, δεν ξεπερνούσε το κατόφλι των 3, του 3% για όλα τα προϊόντα, εκτό από ένα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι για μία κατηγορία, για κάποια συγκεκριμένα ε, ε, ε, ε, προϊόντα ανοξίδου του χάλιβα, η Ινδονησία έχει ξεκινήσει να εξάγει σε μεγάλες ποσότητες. Οπότε είναι σημαντικό για μας να παρακολουθήσουμε το κατά πόσο η Ινδονησία και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες έχουν όντως ξεπεράσει αυτό το όριο του 3%. Και αν ισχύει αυτό, τότε να αποφασίσουμε αν θα τις συμπεριλάβουμε στην, στα μέτρα διασφάλισης ή όχι. Επίσης, να πω ενημερωτικά ότι ε, πολλά μέλη του ΠΟΕ συγκεκριμένα η Τουρκία, η Βραζιλία, η Ταϊβάν και η Ρωσία έχουν κοινοποιήσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση την πρόθεση τους να επιβάλλουν εξισορροπητικά μέτρα για να αποζημιωθούν ε, για την απώλεια εμπορίου που, έχει, λόγω των, που έχουν λόγω των μέτρων που έχουμε επιβάλει. Εμείς είμαστε σε επαφή με αυτά τα μέλη του ΠΟΕ για μας είναι ύψη τη σημασία να διασφαλίσουμε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι ότι βεβαίω οι ρήτρε αυτές διασφάλισης είναι απολύτω νόμιμες σύμφωνα και με τους κανόνες του ΠΟΕ και ότι οι κανόνες του ΠΟΕ επιτρέπουν την επιβολή αποζημιώσεων, αλλά τρία χρόνια μετά την επιβολή των μέτρων διασφάλισης. Οπότε για να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση αποζημίωσης θα πρέπει να φτάσουμε στο 2021. Σίγουρα πάντως δεν θα γίνει τώρα το θα, η συζήτηση αυτή. Είναι σημαντικό λοιπόν να το γνωρίζουν ε, όλοι αυτό. Γιατί η επιβολή των ε, μέτρων διασφάλισης ε, προφανώς δεν είναι ποτέ ανώδυνη, αλλά αποφασίσαμε να το κάνουμε γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν γενικός προς το συμφέρον μας. Και σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Ρινά, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να επανέλθω στο θέμα για την Ινδονησία αναφερθήκατε στο γεγονό ότι η Ινδονησία δεν ήταν χώρα που στοχεύαμε από τα μέτρα διασφάλισης και είναι κάτω 3% αλλά ο κλάδος μας λέει ότι οι εισαγωγές inox και κρύος επεξεργασμένου είναι 18,1 ε, για το πρώτο και 10,1 για το πρώτο και άνω του 3% για το δεύτερο. Υπάρχει πιο συγκεκριμένη πληροφορία από πλευρά ε, ε, επιτροπής Επιτροπή. Μα λέτε ότι για το 18 είναι κάτω 3% ενώ βιομηχανία μα λέει 10,1 παραλαμβάνω για το ανοξίδωτο. Επομένω, ποια είναι τα μεγέθη που έχει η Κομισιόν σχετικά με το 3% και αν περιμένουμε υπερβολικά πολύ, ο κλάδος θα υποφέρει. Μήπως πρέπει να επαναξετάσουμε λοιπόν τα μέτρη διασφάλισης ως προς την Ονδυνησία αντί να περιμένουμε κι άλλο. Ευχαριστώ κύριο Σόλτς. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επιτροπή για τις συγκεκριμένε πληροφορίε. Έχω και εγώ κάποιες πρόσθετες ερωτήσεις. Πρώτον, μπορείτε να μας ενημερώσετε για, το, για την τελευταία συνάντηση του φόρουμ του Χάλιβα του G20. Τι συμφωνήθηκε εκεί. Γιατί θα πρέπει να έχουμε μια συνολική παγκόσμια εικόνα σχετικά με τα του Χάλιβα. Δεύτερον, η αφαίρεση κάποιων, μάλλον η έκπτωση σχετικά με συγκεκριμένες εισαγωγές αμερικανικές μετά τα μέτρα του τμήματος 232, τι σημαίνουν αυτά πιο μακροπρόθεσμα. Έχουμε κάποια προοπτική και σχετικά με, το, με την πρόθεση ανοίγματο διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ, τι θα κάνουμε. Είμαστε σε θέση να άρωμε διασφαλίσεις μάλλον δασμούς που είχαν υποβληθεί υπό το 232. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την εικόνα που μας μετέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι... Δεν θέλω να οδηγώ τη συζήτηση ξανά και ξανά στο Brexit, αλλά τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες συζητούμε πολύ για την Τελωνιακή Ένωση στη χώρα μου και το κατά πόσο θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε πιο αποτελεσματικά εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης την δική μας βιομηχανία και επομένως με μεγάλη ικανοποίηση ακούμε τα μέτρα διασφάλισης για τον Χάλιβα, ιδιαίτερα εν του γεγονότος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πάντοτε πίεζε να έχουμε ισχυρά μέτρα εμπορικής αμήνης εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είχα την ίδια ερώτηση όπως και η κυρία Αρενά για την Ινδονησία. Πόσο γρήγορα μπορούμε να κάνουμε κάποιες προσαρμογές δεδομένων των μεγεθών που μας δίνει ο κλάδος. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια πραγματική δοκιμή του κατά πόσον το πρότυπο ΟΑΣΑ είναι αποτελεσματικό ώστε να αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η προσέγγιση G20 που χρησιμοποιεί τον ΟΑΣΑ γραμματιακά μας οδηγεί σε αποτελεσματική οδό. Μου φάνηκε εκπληκτικό το σχόλιο ότι τα τρία έτη είναι υπερβολικά πολλά, αλλά δεν φαίνεται να έχει αλλάξει τίποτα στην αμερικανική στάση. Τελικά τα τρία χρόνια είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πραγματικά. Έχουμε κάποια ένδειξη ότι οι Αμερικανοί θα αλλάξουν στάση. Υπάρχει κάτι που μας έχει πείσει ότι δεν πρέπει να αντιδράσουμε στα μονομερή αμερικανικά μέτρα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Λεοπόλντο, επομένω από πλευρά μα, αυτά είναι τα ερωτήματα. Αναφερθήκατε στην χρήση κάποιων ποσοστώσεων από κάποιες χώρες άμεσα. Α, ζητώ συγγνώμη, ο κύριος Πάκετ. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα μιλήσω Ολλανδικά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. το κλείσιμο της αμερικανικής αγοράς ε, και η, ε, το εξαιρετικά μεγάλο αποθεματικό στην Ασία, ιδιαίτερα στην Ινδονησία, οδήγησαν σε ισχυρή πίεση προς τον ε, ευρωπαϊκό χάλιβα και ιδιαίτερα οι τιμές του νικελίου που έχουν άμεσο αντίκτυπο επί της τιμής των προϊόντων χάλιβα. Αυτά είναι άμεση απόρρια της Ινδονησίας και το αυξημένο της δυναμικό οφείλεται στην τιμή πρώτων υλών όπως το νικέλιο που είναι πολύ χαμηλότερο από την επίσημη τιμή που δίδεται στην αγορά πρώτων υλών. Και εδώ έχει στρεβλωθεί η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Από πλευρά ACR λοιπόν ζητούμε από την Κομισιόν να καλύψει την Ινδονησία στα μέτρα που μας ανακοίνωσε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ε, επανέρχομαι στο δικό μου ερώτημα. Ακούμε ότι κάποιες χώρες χρησιμοποιούν την ποσόστοσή τους αμέσως. Ποια είναι η συνέπεια. Μήπως πρέπει να επανέλθουμε σε τριμηνιές ποσοστώσεις ώστε να υπάρχει ένα περιθώριο για το σύνολο του έτους. Ή μήπω πρέπει να πάμε σε κατά δασμολογική ποσόστοση ή να περιορίσουμε τα περιθώρια δυναμικού συγκεκριμένων χωρών και συγκεκριμένα για το 5% αύξηση την χαλάρωση, λέει ο πρόεδρος. Μήπως είναι υπερβολικό αυτό σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά του Χάλιβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα το ξαναδείτε το της αύξησης 5%. Γιατί η αγορά του Χάλιβα είναι εξαιρετικά εύθραυστη και με τις τελευταίες προβολές ανάπτυξης που έχουμε τα πράγματα δεν φαίνονται καθόλου ελπιδοφόρα. Μήπως πρέπει να ξαναδείτε το 5%. Thank Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω από το θέμα της Ινδονησίας. Η εφαρμογή τέτοιων μέτρων προστατευτικών πάντοτε γίνεται με βάση μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει και μια κατά αντιπαράσταση ε, συζήτηση μεταξύ των μερών, των ενδιαφερόμενων και βασίζεται και σε δεδομένα. Γιατί σε έρευνες λοιπόν αυτές χρησιμοποιήσαμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία τα οποία κάλυπταν μέχρι και την περίοδο του Ιουνίου 2018. Μέχρι τότε και αυτό μας το έχει επιβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Χάλιβα με τις επιστολές τους. Η Ινδονησία μέχρι τότε δεν είχε ξεπεράσει το 3%. Φαίνεται ότι το ξεπέρασαν περίπου στα μέσα του 2018. Και σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδει η Eurostat, ε, ε, είχαμε τα τελευταία στοιχεία πριν από τρεις εβδομάδες περίπου. Αυτό σημαίνει ότι έτσι μπορούμε να έχουμε ε, στοιχεία για να κάνουμε ένα σωστό υπολογισμό των εισαγωγών. Αλλά επίσης είναι σημαντικό να δίνουμε τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που τους αφορά αυτό το ποσοστό, αυτές τις εισαγωγές, να έχουν τη δυνατότητα να ε, παρεμβαίνουν. Επομένως δεν είναι απλώς ένα ζήτημα ε, μαθηματικού υπολογισμού. Είναι μια διαδικασία εξέτασης. Και για να ε, διεξαχθεί αυτή η διαδικασία εξέταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια σειρά από βήματα. Πολλοί θεωρούν ότι είναι υπερβολικά αυτά τα βήματα, αλλά ε, το θεωρούμε απαραίτητο για λόγους ασφαλεία δικαίου, για λόγους ε, ορθή διαδικασία. Πρέπει να επιτρέψουμε σε όλου του ενδιαφερόμενου να εκφράσουν τι θέσει του. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνει και η αναθεώρηση. Και για κάποια από αυτά τα προστατευτικά μέτρα ε, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι επίγουσα. Γι' αυτό ε, εξετάζουμε το ενδεχόμενο η αναθεώρηση να γίνει πιο νωρίς από τον Ιούλιο, από δηλαδή τη στιγμή που είχαμε αρχικά αναφέρει. Επομένως δεν είναι έλλειψη στοιχείων, το ζήτημα είναι να ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία. Δεν ε, είχα τη δυνατότητα να διαβάσω ακόμα, ή να ενημερωθώ για το τι έγινε στο φόρουμ Χάλιβα, και μπορώ να, δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή, μπορώ να επανέλθω. Για το ερώτημα που μου θέσατε για την κατάσταση της αγοράς χάλιβα, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Θεωρούμε ότι είναι παράνομα στο πλαίσιο των κανόνων του ΠΟΕ τα μέτρα που έλαβαν οι Ηνωμένε Πολιτείες με βάση το, το, το, ε, την νότητα 232 ε, της νομοθεσίας τους. Ε, εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι η λύση είναι να τα αποσύρουν, να τα καταργήσουν. Όταν συμβεί αυτό, τότε πια ο κίνδυνος ε, για την εκτροπές των ροών από, από τρίτες χώρες που εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειωθεί. Και έτσι λοιπόν προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε να πιέσουμε τι ΗΠΑ να αποσύρουν αυτά τα μέτρα. Το πρώτο βήμα θα πρέπει να γίνει όμω από την πλευρά των ΗΠΑ. Πολιτείων. συζητούσαμε αυτά τα θέματα πριν από 2-3 χρόνια. Είχα φέρει τα εξή. Με βάση τους κανόνες του ΠΟΕ, όταν έχουμε τέτοια προστατευτικά μέτρα τα οποία ε, ξεπερνάνε τα τρία χρόνια, ξεκινάει και η δυνατότητα ε, κάποιο να ζητήσει αποζημίωση. Όπω εδώ έχουμε την περίπτωση αυτών των προστατευτικών μέτρων που έχουν δημιουργήσει ζημιά στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Χάλιβα. Πέρα όμω από ε, αυτά τα μέτρα, τα προστατευτικά και τα περιοριστικά του εμπορίου που βλέπουμε να επιβάλλονται σε διάφορα μέρη του κόσμου, συνεχίζει να είναι πολύ δυναμική η αγορά χάλιβα παγκοσμίω. Επομένω, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούσε να παγώσει την αγορά τη, την κατάσταση στην αγορά τη μετά τη Δευτέρα Φεβρουαρίου του 2018, αυτό δεν θα ήταν, και για τρία χρόνια, αυτό δεν θα ήταν και πολύ έξυπνο. Γι' αυτό προτείνουμε να γίνεται μια επαναξιολόγηση, παρά το γεγονό ότι δεν προβλέπεται αυτό ούτε στη δικιά μα νομοθεσία ούτε στου κανόνε του ΠΟΕ, αλλά το χρειαζόμαστε, θεωρούμε, για να, ε, λαμβάνουμε υπόψη μα τη δυναμική κατάσταση τη εξελίξη στην αγορά. Και με αυτά που γίνονται με την Ινδονησία ε, θεωρώ ότι επιβεβαιώνεται αυτή η επιλογή, ότι ήταν σωστή επιλογή. Ε, έχουμε λάβει γνώση και της επιστολής του Πρόεδρου Ταγιάννη προς τον Πρόεδρο Γιούνκερ που ζητάει να συμπεριληφθεί και η Ινδονησία στα μέτρα. Έχουμε, γνώση, έχουμε λάβει γνώση λοιπόν. Ε, για το ερώτημα που μου θέσατε τώρα σε σχέση με τις ποσοστώσεις, η θέση μας είναι να έχουμε και γενικές ποσοστώσεις και ποσοστώσεις συγκεκριμένα σαν χώρα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν ένα ή δύο ε, χώρες οι οποίες να είναι πολύ ανταγωνιστικές και με αυτόν τον τρόπο να κατακτήσουν όλη την αγορά όπου ε, σε κάποια προϊόντα όπως κάποιες ράβδους ας πούμε όπου υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός ε, εάν κρατατήσουμε τον ίδιο, την ίδια ποσόστοση για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω αν θα, τον, θα την κάλυπτε πλήρως η Τουρκία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το να έχουμε και συγκεκριμένες ποσοστάσεις ανά χώρα μας επιτρέπει να περιορίζουμε τις εισαγωγές από αυτή τη συγκεκριμένη χώρα. Τώρα γνωρίζουμε ότι σε πολλούς από τους εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει υπερπαραγωγή, η δυναμικό για υπερπαραγωγή, όχι μόνο στην Κίνα, και για, σε πολλού, πολλούς από αυτούς ο στόχος είναι να κάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες εξαγωγές. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν εάν υπάρχουν ενδείξεις που να μας λένε ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή αυτών των ποσοστώσεων ή να υιοθετήσουμε την ε, γενική ποσόστοση λίγο πιο νωρίς από το τελευταίο τρίμηνο του έτους ε, κτλ. Όμως η βασική μας θέση είναι ότι αυτό το σύστημα είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατευτούμε από κερδοσκοπικές επιθέσεις από συγκεκριμένους προμηθευτές. Τώρα, κατά τα άλλα, ο Χάλεβας πράγματι ακολουθεί πολύ στενά της ε, τάσης οικονομικής ε, ανάπτυξης και πράγματι δεν έχουμε μια ε, ανάπτυξη του 5% στην Ευρώπη. Επομένως αντιλαμβανόμαστε και συμφωνούμε μαζί σας ότι η αύξηση κατά 5% είναι κάπως μεγάλη. Όμως ταυτόχρονα θα θέλαμε η εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης, των προστατευτικών μέτρων θα πρέπει να γίνει σταδιακά. μην ξεχνάτε ότι την προηγούμενη φορά που αναλάβαμε τέτοια μέτρα η αύξηση ήταν 10%. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε μία μέση οδό ανάμεσα στο, 10, στο 0% και το 10% και καταλήξαμε στο 5%. Όμως αυτό δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας ε, ε, επιστημονικής μεθόδου, είναι απλώς ένα συμβιβασμός. Κάτι τελευταίο. για να υιοθετηθούν τέτοια μέτρα προστατευτικά χρειάζεται στο επίπεδο της επιτροπολογίας να υιοθετηθούν, να εγκριθούν από τα κράτη-μέλη με αυξημένη πλειοψηφία. Και γνωρίζετε ότι υπάρχουν διεστάμενες απόψεις στα κράτη-μέλη, ε, γιατί σε κάποια κράτη-μέλη όλος ο τομέας, όλος ο κλάδος αυτός της οικονομίας εξαρτάται από τις εισαγωγές Επομένως προσπαθούμε, αν δεν μπορούμε να του έχουμε τουλάχιστον όλους ικανοποιημένους, τουλάχιστον να είναι όλοι εξίσου, όλοι εξίσου ανήσυχοι, λιγότερο ικανοποιημένοι. Κύριε Σούλτς, εγώ θα ήθελα να σας να επανέλθω στο ζήτημα της συντονισίας. Ζητούμε, για παράδειγμα, από, τους, ε, από το τομέα των πετρελαϊκών ε, να μειώσει την παραγωγή για λόγους ε, περιβαλλοντικούς. Βλέποντας λοιπόν την κατάσταση της οικονομίας και τη διαφοροποίηση που έχει στην οικονομία της, δεν θα ήταν σκόπιμο να δούμε τι είναι αυτό που τους επιτρέπει. Και μήπως ο Χάλιβας είναι πιο σημαντικός και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης Μήπως λοιπόν υπάρχουν κάποια προϊόντα στα οποία θα έπρεπε να επιβάλλει μέτρα η Επιτροπή. Απάντηση. Η εξέταση περιορίζεται στον αγορά του χάλιβα. Δεν εξετάζουμε άλλες αγορές, άλλους κλάδους της οικονομίας. Πολιτικής χρειάζεται η ερώτηση, διπλωματικής η απάντηση. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε στο σημείο 10. Έκθεση, ετήσια έκθεση για τις ε, ε, δραστηριότητες ε, της εμπορικής άμυνας και τη χρήση μέσων εμπορικής άμυνας. Λεοπόλτο και πάλι έχεις το λόγο. Λοιπόν, ανάμεσα στα διάφορα αποτελέσματα του ε, εξυγχρονισμού των μέσων εμπορικής άμυνας, Υπήρχε μια επιθυμία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, υπάρχ, να είναι λίγο πιο λεπτομερείς ε, και μακροσκελής οι ε, ε, εκθέσεις για τις δραστηριότητες αυτές. Αυτή λοιπόν είναι η έκθεση που έχει οθετήσει εδώ και λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια και να σας παρουσιάσουμε πριν από, τη το τέλος της θητείας την έκθεση αυτή. Στο παρελθόν οι εκθέσεις αυτές δημοσιεύονταν το, στο δεύτερο εξάμενο του έτους, αλλά θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό γιατί στα πλαίσια τούτης της ε, θητείας του Κοινοβουλίου ε, είχαμε τις περισσότερες πολιτικές συζητήσεις για την εμπορική άμυνα και ε, αποφασίσαμε να, αποφασίσουμε αυτή, να δημοσιεύσουμε αυτή την έκθεση για να καλύψουμε δύο πράγματα. Να δούμε δηλαδή τι χρειάζεται από το νέο εξυγχρονισμένο κανονισμό. Έχουμε δηλαδή μια αναφορά των δραστηριοτήτων του 2018, αλλά θεωρήσαμε ότι είναι και σημαντικό να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ε, ε, σύνταξης της νομοθεσίας αυτής και κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Γιούγκερ. Ε, κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών των πέντε χρόνων ε, ήταν πραγματικά πολλές οι προκλήσεις και οι οικονομικές και πολιτικές που αντιμετωπίσαμε. Χρησιμοποίησαμε τα εργαλεία εμπορική άμυνα με αποτελεσματικό και στεναρό τρόπο αλλά και ισορροπημένο για να μπορέσουμε να ε, επιτύχουμε τους στόχους που είχαμε υποσχεθεί και να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τα διαθέσιμα μέσα. Το βασικό αποτέλεσμα είναι ότι θεωρούμε ότι έχουμε ε, εξασφαλίσει, προστατεύσει τις, ε, βιομηχα... τις βιομηχανικές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τα μέτρα που επέβαλε η Επιτροπή Juncker μέχρι στιγμής έχουν επιτρέψει να διατηρήσουμε πάνω από 124.000 άμεσες θέσεις εργασίας στον κλάδο της βιομηχανίας. Στο τέλος του 2018, αν δείτε τα μέτρα που έχουν επιβληθεί, θεωρούμε ότι προστατεύσαμε 320.000 θέσεις εργασίας στον βιομηχανικό κλάδο από τον αθέμητο ανταγωνισμό. Πώ δημιουργούμε θέσει εργασία. Βλέπουμε ότι τα μέτρα αυτά του anti-dumping και, και τα αντίθετα με τις επιδοτήσεις έχουν να κάνουν με τις βασικές τιμές εισαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα μας είχαν ε, σημαντικό αντίκτυπο ε, λόγω της, ε, ακριβώς επειδή μείωσαν περίπου 90% σε κάποιες πρόσφατες περιπτώσεις, στις εισαγωγές αυτές, αλλά επειδή είναι πολύ περίπλοκη η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε προϊόν που εισάγεται χρησιμοποιείται και άντι, θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη να επιβάλλει με το μικρότερο δυνατό κόστος για αυτήν αυτά τα μέτρα. Και επίσης είπαμε ότι τα, μέτρα, τα μέσα μέτρα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι χαμηλότερα από τα μέσα μέτρα που επιβάλλουν άλλοι εμποριακοί εταίροι, όπως ας πούμε η ΕΠΑ. Αλλά αυτό το χαμηλότερο επίπεδο δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος ε, στα, στις εισαγωγές. Επίσης, τονίζουμε την, αντιμετώπιση, την προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τις επιδοτήσεις ε, μέσω νέων 25 ερευνών που κάνουμε και από το 2014-2018 καταγράφουμε και στο staff working document που θα έρθει κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι έχουμε διαπιστώσει από τις διάφορες έρευνες που κάνουμε. Να προσθέσω ότι άλλο ένα σημείο που μας επιτρέπει να δούμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος είναι να δούμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά τις, ε, τις, ε, έχουν εκπνεύσει, ε, όσες έρευνες έχουν εκπνεύσει και αναθεωρήσεις. Επίσης, η έκθεση μας δείχνει το τι έχουμε κάνει, μας κάνει έναν απολογισμό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να προλάβουμε την επιβολή παράνομων ε, μέτρων εμπορική άμυνα ε, έναντι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, καταγράφονται αρκετά παραδείγματα μεταξύ πάνω από 70 παρεμβάσεων που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρους των Ευρωπαίων παραγωγών σε τρίτες χώρες. Βεβαίως η έκθεση αυτή τονίζει και την πολύ σημαντική νομοθετική μεταρρύθμιση που έχει γίνει κατά τη διάρκεια του της ε, εντολής, της θητείας και αναφερόμαστε και σε κάτι που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το θέμα των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών πτυχών στις έρευνες αυτές της εμπορικής άμυνας. Ε, ακριβώς επειδή ο εξοχωρισμός της εμπορικής άμυνας ξεκίνησε και τέθησε ισχύ μόλις το 2018, στα τέλη του 2018 δεν είχαμε επαρκέ υλικό για να μπορέσουμε να αναφέρουμε το τι έχουμε κάνει, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε την έκθεση του 2019. Αλλά θέλω να τονίσω ότι ήδη έχουμε έναν μεγάλο αριθμό ερευνών που έχουν ξεκινήσει σύμφωνα με τους νέους κανόνες και βεβαίως σε όλες αυτές τις ε, έρευνες τίθεται πάντα η πτυχή των κοινωνικών και ε, περιβαλλοντικών προτύπων. Αυτά λοιπόν είναι το ζουμί της υπόθεσης. Να προσθέσω ένα τελευταίο σημείο που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Καταγράφουμε και τις ε, επιτόπου επισκέψεις που κάνουμε για τις παληθεύσεις ε, που κάναμε κατά τη διάρκεια του 2018 και οι ε, επισκέψεις αυτές που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε σε βάθος την πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και έφτασαν τις 1978 εργατοημέρες για τους υπαλλήλους της Κομισιόν να πάνε είτε εντό είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να επισκεφθούν επιτόπου και να επιληθεύσουν τις ε, πληροφορίες που έχουμε λάβει για να είναι σίγουροι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουμε για να επιβάλλουμε μέτρα βασίζονται στα πιο ακριβή στοιχεία. Σταματώ εδώ, Πρόεδρε, και αν έχετε ερωτήσεις, ευχαρίστως να σας απαντήσω. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και για την εξήγηση. Ήθελα δύο ερωτήματα να σας υποβάλω. Σχετικά με τα νέα μέσα εμπορικής αμήνης. Τι πρόβολες έχετε σχετικά με το IPI για τις δημόσιες προμήθειες. Η έκθεση ήταν σαφή σχετικά με την ανάγκη να χρησιμοποιούμε, να χρησιμοποιήσουμε μάλλον το μέσο αυτό πριν το τέλος του έτους. Αλλά στο, από το Συμβούλιο έχουμε πολύ πιο ανάμεικτες ενδείξεις. Εσείς τι λέτε. Τώρα για τις ρήτρε διασφάλισης δεν ήθελα τα μέτρα διασφάλισης δεν ήθελα να κάνω το, το ερώτημα στην προηγούμενη συζήτηση γιατί δεν ασχολούμαι γιατί δεν ήξερα τις λεπτομέρειες του Χάλιβα αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς βιομηχανίας που συνδέονται με τα γεωργικά ή με συγκεκριμένα βιομηχανικά προϊόντα παραδοσιακών παραγωγών όπου δυσκολεύονται να ξεκινήσουν μια διαδικασία με την απαραίτητη αν θέλετε αποφασιστικότητα. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στην περιφέρεια της Βαλένθια σχετικά με την εισαγωγή ε, ε, εσπεριδοειδών από χώρες της Αφρικής αλλά όχι μόνο. Εσείς έχετε σκεφτεί μια επανεξέταση του πώς μπορεί να αντιδράσει κανείς αυτοματοποιημένα αν θέλετε για να αντιμετωπίσει τέτοιες εμπορικές εξελίξεις ή θα είναι το μέτρο διασφάλισης το μόνο στο οποίο θα θα σε αντίστοιχη περίπτωση. Ο κύριος Σόλτς, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ και για την ενημέρωση. Πρόσθετο ερώτημα. Με την νέα νομοθεσία που έχουμε για τα μέτρα αντι-dumping κατά των επιδοτήσεων έχουμε εισαγάγει και την ε, δυνατότητα δοκιμής του κατά πόσον υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ. Σε ποιο βαθμό αυτό ε, υλοποιείται πλήρως, εφαρμόζεται ώστε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Επίσης είχαμε την έκθεση για την Κίνα σχετικά με τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποιο βαθμό προσχεδιάζετε, έχετε την πρόθεση να υποβάλλετε και άλλες εκθέσεις ανά χώρα. Γιατί νομίζω ότι δεν πρόκειται μόνο για την Κίνα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή προετοιμάζετε κάποια άλλη έκθεση, αλλά νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία είναι αληθή και για το Βιετνάμ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και από πλευράς μου δύο ερωτήματα. σχετικά με την εναλλακτική μέθοδο υπολογισμού. Είχαμε μια δύσκολη συζήτηση για το θέμα αυτό με την Κίνα και ασκήθηκε και πίεση επί της εναλλακτικής αυτής μεθόδου. Τώρα πώς έχει το πράγμα. Είναι λευκός ή μαύρος ο καπνός. τι προοπτικές υπάρχουν εδώ για το νομοθέτημα αυτό. Δεύτερον, για τα συγκεκριμέ... μάλλον σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο για τα μέτρα αντι-dumping και την ε, ταξινόμηση συγκεκριμένων προϊόντων. Τι δυνατότητες έχουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να υπρασπιστούν θέση τους. Είχαμε πολλές συζητήσεις για την σωστή ταξινόμηση και την πραγματική πρόσβαση που έχει κανείς για να συνομιλήσει με την ε, Κομισιόν. Υπάρχουν νικητές και χαμένοι στα παιχνίδια αυτά και πολύ συχνά οι χαμένοι είναι οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις. υπάρχει για αυτές πραγματική δυνατότητα, επαναλαμβάνω, να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Ευχαριστώ, λέει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Για το μέσο διεθνών προμηθειών, το οποίο εκφεύγει τις διατάξεις, αλλά έστω η Κομισιόν υιοθέτησε την ανακοίνωση για την Κίνα, στην οποία υπογραμμίσαμε έτη το διεθνές αυτό μέσο για τις δημόσιες προμήθειες. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Ιδιαίτερα συμβούλιο, το Συμβούλιο μάλλον δεν υπήρξε σε θέση να έχει επίσημη θέση επ' αυτού. Εμείς πάντως επιμένουμε και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο νομοθεσίας που θα ήταν προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσει προκειμένου να αντιμετωπίσει διάφορες απειλές. από τρίτες χώρες συμπεριλαμβανομένης της Κίνας. Και επομένως πραγματικά και θερμά ελπίζουμε οι συνομοθέτες να υιοθετήσουν το μέτρο αυτό, τη διάταξη αυτή, το συντομότερο δυνατό. Για την ε, εφαρμογή τη λειτουργία του συστήματος. Τα μέτρα διασφάλισης είναι λίγο διαφορετικά από τα μέτρα anti-dumping. Ένα έρευνα επιμέτρου διασφάλισης μπορεί να ζητηθεί από κράτος μέλος και όχι απλώς από τον κλάδο, από τη βιομηχανία γιατί κατά τα άλλα δρούμε κυρίως επί τη βάση καταγγελιών που λαμβάνουμε από τη βιομηχανία γιατί είναι σημαντικό να έχουμε καταγγελίες γιατί προκειμένου να ξεκινήσουμε μια έρευνα χρειαζόμαστε αποδείξεις, ενδείξεις για τις τιμές και τις συνθήκες της βιομηχανίας και μόνο η βιομηχανία είναι σε θέση να μας πει τι ακριβώς, πώς ακριβώς έχει η οικονομική της κατάσταση λέει ο ομιλητής. Στην Κομισιόν έχουμε μια υπηρεσία που ονομάζουμε Γραφείο Παραπώνων. Προς το συμφέρον των πολιτών, λέει ο ομιλητής, και της βιομηχανίας. Και εκεί αναμένουμε επαφές από τη βιομηχανία για να δούμε σε ποιο μέτρο μπορούμε να εφαρμόσουμε το μέτρο αυτό και εφόσον δούμε ότι υπάρχει συνεργασία, είμαστε απόλυτο έτοιμοι να προχωρήσουμε. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα. Ίσως συλλογικά πρέπει να προωθήσουμε λίγο περισσότερο τα μέσα αυτά. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις κράτη-μέλη, η βιομηχανία, η εθνική του κάθε κράτους μέλους, θα τα γνωρίζει αυτά. Είναι αλήθεια ότι η τάση είναι να χρησιμοποιούνται περισσότερο τα μέτρα αυτά από τα κονζόρτια, για να το πούμε έτσι, που εδράζονται στις Βρυξέλλες ή που έχουν παρουσία στις Βρυξέλλες. Είναι αλήθεια αυτό. Κάνουμε μια προσπάθεια στα κράτη-μέλη να παρουσιάσουμε τα μέτρα. Έχουμε ζητήσει από τους εκπροσώπους των κρατών μελών στην Επιτροπή Εμπορικής Αμήνης να διοργανωθούν συναντήσεις όχι μόνο με τις διοικήσεις αλλά με τους εκπροσώπους βιομηχανία και τους κοινωνικούς εταίρους. Είχαμε μια τέτοια συνάντηση πριν από δύο εβδομάδες στην Αυστρία, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όπου προσήλθαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και είμαστε απολύτως διαθέσιμοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή. Τώρα αν μπορώ να πάω στο δεύτερο ερώτημα από την κυρία Λάνγκε η ιστοσελίδα της Επιτροπής έχει έναν οδηγό καταγγελιών και έναν οδηγό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το πιο σημαντικό είναι να εκφράζονται οι ενδιαφερόμενοι, να έρχονται σε επαφή. Ποτέ δεν έχουμε αρνηθεί συνάντηση για να συζητήσουμε συγκεκριμένο πρόβλημα. Έχουμε μέτρα που αφορούν πολύ συγκεκριμένα τον κλάδο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων το ότι είναι κανείς μη μη ε δεν είναι από μόνο του τροχοπέδι. Τροχοπέδι είναι η έλλειψη μιας κάποιας οργάνωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ δεν καλούμαστε να προστατεύσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, αλλά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ο συνεταιρισμός, για να το πω έτσι, χρειάζεται η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των επιχειρήσεων. Πάντως με μεγάλη χαρά συναντόμαστε με τους εκπροσώπους βιομηχανίας για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα κατά πόσον υφίστανται οι συνθήκες για να εκκινήσει η έρευνα και ότι αυτές είναι περιοριστικές είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να είναι και αξιόπιστο. Και αυτό είναι σημαντικό. Για τα πρότυπα τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά θα θυμάστε ίσως του τριμε, τους τριμερείς διαλόγους, οποίους τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι το συμβαστικό κείμενο ήταν λίγο ή πολύ το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Καθότι ο ΠΟΕ δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα περιβαλλοντικού ή κοινωνικού dumping καθεαυτά ως φαινόμενα, αλλά κάτι εισήγαμε ως, ως περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Αυτά τα βλέπουμε στις έρευνές μας και τα λαμβάνουμε υπόψη μας σχετικά π.χ. με τις κατάλληλες τρίτες χώρες για την εναλλακτική μέθοδο υπολογισμού για το dumping σχετικά με τις ε, τιμές που θα πρέπει να υποβάλλονται υπό τον εξυγχρονισμένο κώδικα τιμολόγησης για τις δίκαιες τιμές και με τις νέους κανόνες έχουμε κατευθυντηρές γραμμές για τα θέματα αυτά. Αλλά αυτό είναι το μέγιστο, ο, το, ο μέγιστος βαθμός στον οποίο μπορούμε να κινητοποιηθούμε για τους κανόνες των τρίτων χωρών. Εμείς λαμβάνουμε τις χώρες κατά αύξοντα αριθμό των μέτρων που έχουν επιβληθεί εναντίον τους. Η, Ρωσ... Κίνα είναι στην πρώτη θέση, η Ρωσία στη δεύτερη εξού και ετοιμάζουμε έκθεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη Ρωσία. Είναι δύσκολο να σας δώσω ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα υποβληθεί η έκθεση αυτή, αλλά φαντάζομαι ότι κάποιους μήνες ακόμα θα χρειαστούμε. Όταν θα έχουμε ολοκληρώσει την έκθεση για τη Ρωσία θα δούμε κατά πόσο χρειάζεται να συνεχίσουμε με εκθέσεις και για άλλες τρίτες χώρες, αλλά θα εξαρτηθεί πολύ από τις χώρες τις οποίες προκύπτουν στην καθημερινή μας δουλειά. Τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι καμία έρευνα που να έχει κινήσει κατά του Βιετνάμ, να σας πω. Για τον νέο υπολογισμό για το ντάμπινγκ, πράγματι η Κίνα συμφώνησε στη σύσταση ενός πάνελ για το σύνολο της νομοθεσίας, το οποίο πάνελ εξετάζει τα διάφορα στοιχεία που του έχουν υποβληθεί. Ε, εύχομαι και ελπίζω ότι το πάνελ θα μπορέσει να υποβάλει μια έκθεση και ότι θα τοποθετηθεί υπέρ των σημείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Thanks και εμείς ευχαριστούμε. Θέλεμε θέλαμε όμως να μας δώσετε λίγες περισσότερες πληροφορίες. Τι πιστεύετε, αυτή η πίεση προς την Κίνα α, οδηγεί σε κάποια, αλλαγή της νομοθεσίας και τα λοιπά. Απάντηση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι γνωρίζω ότι η Κίνα δεν, είναι, δεν τη χαροποιούν οι τα μέτρα που έχουμε λάβει για την προστασία του εμπορίου μας και επίσης θεωρούν ότι η μελακλική μέθοδος υπολογισμού ε, εισάγει διακρίσεις εναντίον τους. Βεβαίως διαφωνούμε εμείς με αυτή την αξιολόγηση. Ε, το, δεν θα έλεγα ότι το ζήτημα τους, ε, αυτών των μέτρων είναι ένα θέμα το οποίο να μας απασχολεί συνέχεια στις επαφές με την Κίνα. Είναι ένα σημαντικό θέμα στις σχέσεις μας με την Κίνα. Όμως, όπως έλεγα, έχουμε αυτά τα εργαλεία, τα εφαρμόζουμε και θεωρούμε ότι τα εφαρμόζουμε σεβόμενοι πλήρως τους κανόνες του ΠΟΕ. Απλώς κάνουμε, ασκούμε τα δικαιώματα που έχουμε με βάση τους κανόνες του ΠΟΕ. Τώρα, για να απαντήσω στην ερώτηση σας, βεβαίως δεν είναι χαρούμενη η Κίνα. Σας ευχαριστούμε. Έτσι έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση για το σημείο 10. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών πριν να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες.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 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Πάμε στο σημείο 11 της μερίσιας διάταξης. Η ψηφοφορία είναι η τελευταία ψηφοφορία της Επιτροπής μας για αυτή τη θητεία. Πρόκειται για την Διεθνή Συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές. Ε, μία είναι η ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε όλοι τις κάρτες σας μαζί. Τις κάρτες ψηφοφορίας. Πρώτα απ' όλα θα κάνουμε όπως συνήθως έναν έλεγχο. Ψηφίστε για τον έλεγχο. Ωραία, λειτουργεί και στα σας. Τώρα μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία. Και τώρα, η τελευταία μας ψηφοφορία, όπως σας έλεγα, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα So, Σας ευχαριστώ λοιπόν. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 12, ομάδα παρακολούθησης. Είχαμε δύο συνεδριάσεις της ομάδας παρακολούθησης τις τελευταίες εβδομάδες. Η μία έχει σχέση με την Νοτιοανατολική Ασία. Ησυχία παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Και άλλοι. Ας ξεκινήσουμε με την Νότιο-Ανατολική Ασία. Δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο ε, να σας ενημερώσουν Είναι εδώ ο κύριος Κάμπελ. Πού είναι και δεν τον βλέπω. Στο συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, με... ξαφτιάσατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την παρουσία τους. Θα σας ενημερώσω για την ε, συνεδρίαση της ομάδας παρακολούθησης για την Νοτιοανατολική Ασία που προκείται για υποεπιτροπή δική μας. Ε, εστιάσαμε κυρίως για τις εξελίξεις μετά τις 27 ε, Φεβρουαρίου και την εφαρμογή του ε, συμφώνου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο πρέσβης, ο Μοχάμετ Σαντάτ Χωσαΐν, παρευρέθη και τον ευχαριστούμε. Και συζητήσαμε επίσης και για τις εξελίξεις στις 21 Φεβρουαρίου, ε, στις 21 Φεβρουαρίου συζητήσαμε για την ε, τις εξελίξεις στις άλλες περιοχές του Μπαγκλαντές. Μας ανέφεραν διάφορους τομείς, τους οποίους έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά περιορισμένη. Πρώτα απ' όλα, μία από αυτές είναι το ελάχιστο όριο των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η αναθεώρηση του εργατικού δικαίου και αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να περιοριστούν, από την πλευρά μας ότι θα πρέπει να σταματήσουν και να μειωθούν οι περιορισμοί που επιβάλλονται στο, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η, Επιτροπή, η Υπηρεσία μάλλον Εξωτερικής Δράσης προσπάθησε να μας δώσει και την άλλη πλευρά, λαμβάνοντας ότι και μας είπε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση στον Μπαγκλαντές και την πολύ μεγάλη ε, εισρωή προσφύγων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε είχε τη θέση ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τον Μπαγκλαντέ να ανταποκριθεί σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των συζητήσεων, ενημερωθήκαμε ότι το 70% ε, του χρόνου των ε, Υπουργείων των Αρμόδιων στο Μπαγκλαντές θα ασχοληθεί, ε, αναγκάζεται να ασχολείται με την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, το οποίο περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες της κυβέρνησης να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο. Τώρα όσον αφορά τους επιθεωρητές εργασίας, ενημερωθήκαμε ότι γίνεται μια διαπραγμάτευση αυτόν τον καιρό με την, ε, το Διεθνή Οργανισμό Εργασία για τι διαδικασίε τι σχετικέ και σε σχέση με τον τομέα της κλώστου υφαντουργίας διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασκήσει πίεση και μας ενημέρωσε η Επιτροπή ότι θα ξεκινήσει διάλογο και επικοινωνία με, τους άλλους, με, με τις ε, επιχειρήσεις του, του κλάδου και με τους ενδιαφερόμενους του κλάδου. Πρόκειται για μια συζήτηση η οποία έχει κρατήσει, έχει ξεκινήσει πριν από 7-8 χρόνια. Ε, πριν από 5 χρόνια είχα, ήταν έντονες οι πιέσεις. Μας έλεγαν οι α, επιχειρήσεις ότι κάτι θα έπρεπε να γίνει για τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι τιμές. Δεν έχει συμβεί όμως κάποια εξέλιξη και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αρχίσει να αξιοποιεί τους, τις μεθόδους πίεσης που έχουμε έτσι ώστε να μην μειώνονται συνέχεια οι τιμές, αλλά να μπορεί να δημιουργηθεί και κάποιο περιθώριο κέρδους για αυτές τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να επανεπενδύσουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν και που και εμείς θα θέλαμε να αντιμετωπίσουν. Ναι. Συζητήθηκε επίσης η σχέση των, ε, του Μπαγκλαντές των προεθμιθευτών από τον Μπαγκλαντές με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον χώρο της κλωστοϊφαντουργίας και ότι θα πρέπει να, συνεργαστεί αυτή, να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία για την αντιμετώπιση προβλημάτων που χρονίζουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη συζήτηση με τον Μπαγκλαντέ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργατικών δικαιωμάτων. Ε, Αξιοποιώντα το πλαίσιο ε, συνεργασία με τον Περκλεντέ που έχουμε βάσει το πρόγραμμα «Τα πάντα εκτός από όπλα». Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρέσβη του Μπαγκλαντές και την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής τράση για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της θητεία στο πλαίσιο της Επιτροπής παρακολούθηση τη Νοτιοανατολική Ασίας. ευχαριστώ. Ερωτήσεις υπάρχουν για τον Μπαγκλαντές. Όχι. Ωραία, σας ευχαριστούμε και πάλι. Και πάμε στην Ανατολική Αφρική. Ο Χέλμουντ Σόλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, μια γενική εικόνα της τελευταίας συνάντησης της ε, Ομάδας Εποπτείας για την Κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής έγινε για τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανατολική Αφρική μετά από την τελευταία σύνοδο που έγινε την 1η Φεβρουαρίου. Και είδαμε γενικώ τον απολογισμό και τις ε, τελευταίες ε, αλλαγές που έχουν γίνει στην Τανζανία. Συζητήσαμε γενικώ την πολιτική ε, συζήτηση, στην, στην, την πολιτική κατάσταση στην Τανζανία κυρίως και τις διμερείς σχέσεις, κυρίως ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις, την κατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα και επίσης θέλαμε να έχουμε και μια ενημέρωση για το τι γίνεται στο Μπουρούντι, όπου υπάρχουν παρόμοια προβλήματα. Όπω θα θυμάστε, οι συζητήσει, για τις εμπορικές σχέσεις ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανατολικής Αφρικής είχαν ολοκληρωθεί ε, ήδη από το 2014. Είναι μια συμφωνία που γίνεται με περιφέρειες, ε, υπεγράφηκε, και επικυρώθηκε από, όλες τις, από, τα, από όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από τον Νότιο Σουδάν και έπρεπε να, μπει, να τεθεί σε ισχύ. Από τότε βεβαίως μόνο η Κένια και η Ρουάντα έχουν υπογράψει την συμφωνία αυτή. Το Μπουρούντι, η Ουγγάντα, η Τανζανία δεν έχουν υπογράψει ακόμα. Η Τανζανία λέει ότι θέλει περισσότερο χρόνο για να αναλύσει τον αντίκτυπο της συμφωνίας, να μελετήσει τα θέματα που περιλαμβάνει και ίσως αυτό βεβαίω να έχει να κάνει και με τις προκλήσεις που απορρέουν από το, από το Brexit και, γιατί υπάρχουν διάφορες διμερείς σχέσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τανζανία. Το Μπορούντι έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για τι ε, κυρώσει που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουγγάντα έχει αναλάβει το ρόλο του ενδιαμέσου. Στην, ε, ολοκλήρωση, μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας συνόδου υπάρχει μία έκθεση για τα IPAs και λέει ότι ε, οι κοινότητε των Αφρικανικών της Ανατολικής Αφρικής ε, στους επόμενους τέσσερις μήνες θα είναι σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει διασάφηση για κάποια σημαντικά σημεία. Και μετά οι χώρες εταίροι που θέλουν μπορούν να υπογράψουν την συμφωνία. Αλλά μπορούν και να μην την υπογράψουν θα πρέπει να δούμε τι, πώς ε, θα είναι εφικτό να υπάρξει ε, εφαρμογή της EPA ε με τις, μόνο με τις χώρες που είναι διατεθειμένες να υπογράψουν. Αλλά η απάντηση αυτό τελικώς ήταν όχι, δεν γίνεται. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την ε, Κένια. Θα υπάρχει μια ανοιχτή διάταξη. Για τα υπόλοιπα τώρα μέλη της Ανατολικής Αφρικής θα απολαμβάνουν ε, την πρόσβαση στην αγορά και τα όσα απορρέουν από τη συμφωνία όλα εκτός από όπλα. Οπότε προ το παρόν, ω προ αυτό, ε, έχουμε κάποιε εγγύσει. Τώρα, από πολιτική πλευρά, ε, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Τανζανία και με τον Μπορούντι. Από το 2015 υπάρχουν κυρώσει που έχουν επιβληθεί στου πολιτικού του Μπορούντι που επιβεβαιώθηκαν και πέρσι μέχρι τον Οκτώβριο του, 31 Οκτωβρίου του 2019. Για την Τανζανία τώρα, ε, Έχουμε επιδείνωση του πολιτικού κλίματος, υπάρχει όλο και περισσότερη καταπίεση των ε, κομμάτων της αντιπολίτευση και των βουλευτών, ε, τρομοκρατούνται. Ε, υπήρξε ένα διάταγμα για την καταγραφή των ομοφιλοφίλων στην αστυνομία και ενθαρρύνονται δράσεις εναντίον των ομοφιλοφίλων. Ο πρέσβης αντέδρασε και απελάθηκε από την Τανζανία. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ανακάλεσε τον ε, πρέσβη τη και ε, θα αναθεωρήσει τις διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα. Κάποια κράτη-μέλη ήδη έχουν αναστείλει την αναπτυξιακή βοήθεια που στέλνουν. Οπότε έτσι έχουν ξεκινήσει λίγο να αλλάζουν και τα ανάλυση και νοοτροπία και ο πρόεδρος Μαγκουφούλη έχει αποφασίσει να υπογράψει τη συμφωνία εάν η αναπτυξιακή βοήθεια Ξανασυνεχίσει να ρέει προς την Τανζανία. Και επίσης θα προσπαθήσουν να πείσουν και τον Μπουρούντι να υπογράψει, παρόλο που οι κυρώσεις για τον Μπουρούντι εξακολουθούν να είναι σε ισχύ. Γιατί είναι ιδιαίτερο σημαντική η συμφωνία αυτή για την Τανζανία και τώρα είμαστε σε ένα δίλημα Και πρέπει να δούμε ε, τι να κάνουμε με την κριτική στάση που έχουμε για την κατάσταση που επιδεινώνεται στην Τανζανία, να, το, να σταματήσουμε για να ανταλλάξουμε με την υπογραφή της συμφωνίας. Εγώ θα έλεγα όχι. Εμείς ως Επιτροπή ΙΝΤΑ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στα νερά πίσω από τις αρχές μας ε, που διέπουν τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές απορρέουν από τη συνθήκη, και να ενθαρρύνουμε να, είναι το, να τηρηθούν οι αρχές του δίκαιου εμπορίου και αυτό να ε, ενταχθεί στις συνολικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εξωτερικές δράσεις με τις τρίτες χώρες. Αυτά από μένα, Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Δύσκολη κατάσταση. Και οικονομικά και πιο πολύ πολιτικά. Ε, ερωτήσεις υπάρχουν προς τον Χέλμουτ για την Ανατολική Αφρική. Όχι. Ευχαριστώ και τους δύο Η Οι ομάδες εποπτείας, συναδελφοί, είναι πραγματικά πολύ καλό μέσο για να ε, επηρεαστεί η όλη διαδικασία εφαρμογη αλλά και ίδια πραγματεύσεις. Χθε ακούσαμε έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Λέβεν που μα είπε ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία για την ε, ενίσχυση του Κοινοβουλίου και την ενίσχυση τη ε, επίρριά του στην εμπορική πολιτική. Ευχαριστούμε λοιπόν που αναλαμβάνατε αυτά τα καθήκοντα. Σημείο 13. Κίνα. Έχουμε και παρουσίαση PowerPoint. Να κατέβει λίγο η οθόνη, περιμένετε. Ε, φωνάζω λίγο γιατί κάνει λίγο θόρυβο η οθόνη όσο κατεβαίνει. Οπότε να δώσουμε το λόγο στο συνάδελφο για να κάνει την παρουσίαση του. Για να μας εξηγήσει τη νέα στρατηγική για την Κίνα Έχουμε λάβει εδώ και κάποιες εβδομάδες μια κοινοποίηση, μια ανακοίνωση που μας εξέπληξε. Ήταν λίγο πιο αυστηρή η διατύπωση από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Και επίσης δεν ήταν και απολύτως συμμορφούμενη με τη θέση του Κοινοβουλίου. Τη θέση που υιοθετήσαμε πέρσι με εισηγητή τον κύριο Βίνκλερ. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι να το συζητήσουμε, να τη συζητήσουμε αυτή την, το νέο σκεπτικό της Κομισιόν και ο Πίτερ έχει τώρα το καθήκον να μας εξηγήσει πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα εντός της Κομισιόν. Thank Πρόεδρε, Έχω πέντε λεπτά για να εξηγήσω την στρατηγική για την Κίνα. Αυτό είναι πρόκληση από μόνο του. Υπήρξε και το σχετικό θέμα εχθές. Σήμερα θα μιλήσω για την κοινή ανακοίνωση και την προετοιμασία τη Συνόδου. Η οθόνη δεν είναι για μένα, θα είναι για το συνάδελφο που έπεται. Οπότε αφήστε την οθόνη, λέει ο Μίλτης. Λοιπόν, η αφήγηση σχετικά με την Κίνα έχει αλλάξει. Έχουμε περισσότερη υπογράμμιση των απειλών παρά των ευκαιριών. Και τα υφιστάμενα εθνή μέτρα δεν αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο που ακολουθεί τον κρατικό καπιταλισμό και τον οποίο αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερο ως αντίπαλο. η Κίνα θα μπορούσε να φτάσει στο συμπέρασμα σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση των ΠΟΕ να μην αλλάξει το status quo. Η Κίνα όμως πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της αναλόγως προς την σημασία της στην οικονομική και εμπορική και να αντιμετωπίσει την ανισορροπία που δημιουργεί στο διεθνές εμπόριο ιδιαίτερα με τις επιδοτήσεις της κρατικές της. για τις ανισορροπίες της αγοράς, την πρόσβαση στην αγορά, το υπερβολικά μεγάλο αποθεματικό και τα, τους ισότιμους κανόνες παιχνιδιού όταν ανταγωνίζονται οι δικές μας επιχειρήσεις με τις κινέζικες στις δύο αγορές αλλά και σε αγορές τρίτων χώρων. Ακούμε πολλά σχετικά με άνοιγμα και μεταρρύθμιση από Κινέζους ηγέτες. Αν δει κανεί πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει η μεταρρύθμιση του Προέδρου είναι να προσαρμόσει, να κάνει πιο αποτελεσματικές τις δικές της ε, κρατικά επιδοτούμενες επιχειρήσεις στην διεθνή αγορά. Εν ολίγης πρέπει να πιέσουμε, να συνεχίσουμε να πιέζουμε την Κίνα, να αναλάβει μεταρρυθμίσεις και αντιστάθμιση, εξισορρόπηση στι εμπορικέ μας σχέσει. και θα πρέπει να αναλάβουμε και βήματα για να αντιμετωπίσουμε τη στρέβλωση της αγοράς που οφείλεται στις πρακτικές Κίνας. Στις 12 Μαρτίου, μαζί με την ΙΕΔ, υποβάλαμε μια κοινή ανακοίνωση για τις σχέσεις με την Κίνα. Νομίζω ότι αυτή η ανάλυση δεν ήταν εχθρική ή επιθετική, ήταν όμως ακριβής. Ο στόχος της ήταν να διαβάσει σαφή πολιτικά μηνύματα και να προτείνει απτές δράσεις για να εξισορροπηθούν οι σχέσεις μας με την Κίνα. Η ανακοίνωση συνέβαλε στην συζήτηση στο Συμβούλιο της 20ης Δευτέρας Μαρτίου ευρύτερες συζητήσεις όχι ως προπαρασκευή της Συνόδου στο οποίο θα έρθω σε λίγο και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου παρότι δεν εστίαζαν στην Κίνα αποτύπωναν το περιεχόμενο της κοινή ανακοίνωση η οποία συμπεριλαμβάνει 10 σημεία δράσης στο πλαίσιο των συνολικών σχέσεών μας με την Κίνα. Μεγάλο μέρος των μέτρων αυτών σχετίζονται με το εμπόριο. Η δράση 4 αφορά στην εφαρμογή των διμερών συμφωνιών. FTAs με τους ανατολικούς εταίρους, αλλά και τη στατική διασυνδεσιμότητας που σχετίζεται με το εμπόριο. Δράση 5. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες να εξισορροπήσουμε τους κανόνες παιχνιδιού με την Κίνα που δεν είναι ισορροπή αυτή τη στιγμή. Η μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, η επικαιροποίηση των κανόνων στις βιομηχανικές επιδοτήσεις, οι τεχνολογικές μεταφορές, μαζί με μια συνολική πλήρη επενδυτική συμφωνία. Εν ώψη του να την ολοκληρώσουμε του χρόνου. Επίσης, διμερείς συμφωνίες για τις ε, γεωγραφικές προελεύσεις και την ασφάλεια των αερομεταφορών. Δράση 6 για τον περιορισμό του μοθετικού έργου σχετικά με τα μέσα μέτρα δημοσίων προμηθειών που αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται. Δράση 7 επίσης για τις δημόσιες Αναθεώρηση του υφισταμένου ενωσιακού πλαισίου μαζί με την συμμετοχή εξωτερικών συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς. Δράση 8 για την αντιμετώπιση της τρέβλωσης εξωτερικών κρατικών φορέων στην εσωτερική αγορά και το πώς να πληρώσουμε υφιστάμενα κενά στην νομοθεσία μέχρι το τέλος 19 για την αυξανόμενη παρουσία της Κίνας στην εσωτερική αγορά, στις βιομηχανικές επιδοτήσεις π.χ. που παρέχει η Κίνα προς τις επιχειρήσεις της για να εξαγοράσουν ή να συγχωνευτούν με ευρωπαϊκές ή επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στην ευρωπαϊκή αγορά χάρη σε κρατικές επιδοτήσεις από την Κίνα. Δράση 10 για την αποτελεσματική εφαρμογή του πρόσφατου κανονισμού για το screening στο FDI. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η πρόταση της Κομισιόν για τους εξαγωγικούς ελέγχους και για τις αλυσίδες στρατηγικής σημασίας. Για την εφαρμογή τώρα, την υλοποίηση των σημείων αυτών. Κάποιες από τις δραστηριότητες αυτές ήδη τρέχουν, όπως οι διμερείς διαπραγματεύσει που έχουν την Κίνα. Άλλες θα χρειαστούν περισσότερες εσωτερικές διαβουλεύσεις. Πάω τώρα γρήγορα στην σύνοδο της ερχόμενης εβδομάδας, εδώ στι Βρυξέλλες. Θα είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε την δέσμευση της Κίνας σε διάφορες περιοχές, σε διάφορα πεδία και να ασκήσουμε πίεση εφόσον δεν ανταποκριθεί. Επί τη βάση της περισσυνής δήλωσης έχουμε διάφορα σημεία στα οποία δεν έχει Κίνα εκπληρώσει υποχρεώσει της για τις ε, μεταρρυθμίσεις ΠΟΕ για παράδειγμα για τις ε, διαπραγματεύσεις για τις επενδυτικές συμφωνίες και για την υποχώρησή της σχετικά με τις ε, γεωγραφικές προελεύσεις γεωγραφικές ενδείξεις στην κοινή δήλωση της Συνόδου αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα όπως φαντάζεστε με τους Κινέζους. Διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι θα φέρει η Σύνοδος της 9 η Απριλίου. Εργαζόμαστε σκληρά με τους Κινέζους εταίρους να έχουμε μία δήλωση με περιεχόμενο ουσιαστική. Και μαθαίνουμε ότι τα κράτη-μέλη προτιμούν μια δήλωση ουσιαστική και με περιεχόμενο παρά χωρίς περιεχόμενο και μη ουσιαστική λέει ο μιλητής. Και βεβαίως θέλουμε να έχουμε μια ουσιαστική σύνοδο με ένα ουσιαστικό πόρισμα. Και το ουσιαστικό meaningful στα αγγλικά είναι φορτισμένος όρος αυτή τη στιγμή όπως καταλαβαίνετε λέει ο μιλητής αναφερόμενος στο Brexit αλλά έχουμε κάποια σκληρά καρύδια να σπάσουμε με τους Κινέζους, ιδιαίτερα στα εμπορικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, να δώσω τώρα στον εισηγητή μας το λόγο, καταρχάς. Thank you very much, Chairman, and thank you for this. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό, νομίζω, να το επισημάνει κανείς και είναι και προφανές αλλά είναι θετικό που το επισημαίνει και η Επιτροπή. Είναι λοιπόν σημαντικό να δει κανεί ότι τα περισσότερα από αυτά που αναφέρει ως ε, σχετικά στοιχεία της σχέση μας της μελλοντική με την Κίνα έχουν σχέση με το εμπόριο. Γιατί βεβαίως συνεργαζόμαστε με την Κίνα σε πολλούς άλλους τομείς, πολιτικούς, γεωστρατηγικούς, αλλά ε, η ουσία των σχέσεών μας θα πρέπει να είναι οι εμπορικές σχέσεις. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω θα ε, μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη μελλοντική μας σχέση. Όλα είναι σημαντικά. Τα εργαλεία τα αμυντικά ε, του εμπορίου είναι σημαντικά και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις όλων αυτών των εξέλιξεων στην τεχνολογία. Θα χρειαστεί να το εξετάσει αυτό και το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η αντίστοιχη Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, η επόμενη, αλλά επίσης και η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τον Οκτώβριο. Αναφερθήκατε κι εσείς στο IPI πιστεύω, για τις διεθνείς προμήθειες, πιστεύω ότι και εδώ έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά πρέπει να τα δούμε επιτέλους και στην πράξη να εφαρμόζονται. Για τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, συμφωνώ μαζί σας, θα πρέπει να δούμε από την πλευρά των Κινέζων να υλοποιούν κάποιες από τις δεσμεύσεις τους. Εάν ε, με ρωτάτε εμένα ποιο θα έπρεπε να είναι το μήνυμα προς τους συναδέλφους στην Κίνα, προς τους ε, εταίρους μας στην Κίνα, ε, νομίζω ότι το μήνυμα είναι ότι ήρθε η ώρα να υλοποιήσουν αυτά που υπόσχονται, γιατί τα έχουμε επαναλάβει πολλές πολλές φορές. Πρέπει να τα δούμε όμως και στην πράξη, πρέπει να δούμε πρόοδο. Και κάτι που θέλω να καταγράψω ως ιδέα για την επόμενη Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν θέλετε κύριε Πρόεδρε, η κληρονομιά που θα αφήσουμε στην Επιτροπή αυτή είναι ακριβώς αυτή η αυστηρή ε, στάση που εκφράζει ξεκάθαρα τις θέσεις μας. Αυτό είναι ο, η, η, πηξίδα για την επόμενη Επιτροπή. Γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια ε, εξετάσαμε πολύ λάπερη πλοκά ζητήματα. Ε, εγώ είμαι σίγουρος ότι για, το θέμα της Κίνας θα χρειαστούν δύσκολες αποφάσεις τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω εμείς βάλαμε τα θεμέλια για να συνεχίσουμε αποτελεσματικά και ελπίζω η επόμενη Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η επόμενη Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου να είναι ακόμα πιο αποφασιστικές. Κύριος Μπέλντα, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που θα έχω τη δυνατότητα να ε, μιλήσω ως εισηγητής για το ζήτημα των σχέσεων με την ε, Κίνα. Πρόσφατα ε, διάβασα στην Frankfurt Allgemeine ε, κάποιες, ένα δημοσίευμα για την Κίνα, το, η οποία με εντυπωσίασε, μιλούσε για μια σειρά στη γερμανική τηλεόραση τη αστυνομική και παρουσίαζε την Κίνα σαν ε, μια χώρα η οποία έχει φροντίσει να στείλει κατασκόπους παντού σε ολόκληρη την Ευρώπη. οι ε, επενδύσεις από την πλευρά των Κινέζων έχει εκτιμηθεί, λέει, λέει το δημοσίευμα, ότι έχουν δημιουργήσει ε, μια απώλεια της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ για γερμανικές επιχειρήσεις ε, και, όταν τι θα έπρεπε να κάνει κανείς για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Συζητάμε πολύ συχνά λοιπόν το πρόβλημα της Κίνας. Πρόκειται, μας ξεπερνάει το μέγεθος της χώρας και με χαρά διάβασα αυτή την έκθεση που αναλύει την ευρωπαϊκή πολιτική για το διεθνές εμπόριο και που είχε πολύ ενδιαφέρον μάλιστα ότι έλεγε ότι θα πρέπει κανείς να μπει και στην θέση των Κινέζων, να αντιληφθεί την δική τους κοσμοθεωρία, πώς αντιλαμβάνονται τον ε, κόσμο, τη θέση τους σε αυτόν και το εμπόριο γενικότερα. Ε, επίσης αναφέρθηκε ότι δεν θα πρέπει να υποτιμούμε την κατάσταση της την εσωτερική στην Κίνα. Ίσως η χώρα αυτή να μην είναι τόσο σταθερή όσο νομίζουμε. Ε, και επίσης ε, έλεγε η έκθεση ότι θα, δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε εμείς οι Ευρωπαίοι να είμαστε αφελείς απέναντι στο τι συμβαίνει στην Κίνα. Πολλά από αυτά τα στοιχεία λοιπόν με εντυπωσίασαν. οι ειδικοί, πανεπιστημιακοί και άλλοι, λένε ότι θα αναμείνουμε μία ε, υποχώρηση της ανάπτυξης, ε, επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στην Κίνα τα επόμενα 5 με 10 χρόνια. Αυτό βέβαια είναι μια πρόβληψη που βασίζεται σε αναλύσεις. Ωστόσο, είναι σίγουρο ότι αν υπάρχει τέτοια επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξη στην Κίνα, θα δημιουργηθούν κρίσει, οι οποίε θα έχουν επιπτώσει και στο εσωτερικό τη Κίνα αλλά και διεθνώ. Επομένω, εμεί θα πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό το ενδεχόμενο. Και να είμαστε έτοιμοι να ε, να, να ασχοληθούμε ουσιαστικά με το θέμα αυτό. Να, να μην διστάσουμε. Αν έρθουν τέτοιες κρίσεις, αν συμβούν τέτοιες κρίσεις στην κινέζικη οικονομία, είναι σίγουρο ότι θα έχουν επιπτώσεις και στα δικά μας συμφέροντα. Κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε πλέον να μιλούμε για ένα ολοκληρωτικό καθεστώς στην Κίνα. Είμαι ιστορικός, γνωρίζω ότι στο παρελθόν στην Κίνα υπήρχαν, υπήρχε ολοκληρωτικό καθεστώς, αντίστοιχο με εκείνο της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά δεν πιστεύω ότι το σημερινό καθεστώς στην Κίνα μπορεί να το χαρακτηρίζει κανείς ολοκληρωτικό. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό και νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει ποιος είναι ο ρόλος των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο κινέζικο σύστημα, καθώς επίσης και ο ρόλος των κρατικών επιχειρήσεων στο κινέζικο σύστημα. Γνωρίζουμε ότι το, μοντέλο της Κίνας είναι να έχει η κυβέρνηση μια πολύ μεγάλη επιρροή στις επιχειρήσεις, ε, και γνωρίζουμε πως αυτό το αξιοποιούν για να προχωρούν και να εισάγουν και, να, να, να επενδύουν σε αγορές τρίτων χωρών και γνωρίζουμε επίσης πώς αυτό πλήττει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το μεγάλο δυναμικό της Κίνας δημιουργεί προβλήματα στις, στο διεθνές εμπόριο. Όμως πρέπει να δούμε και την εσωτερική οικονομία στην ε, Κίνα Έχουμε επίσης το ζήτημα της τεχνολογίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, δηλαδή θέλουμε οι κινέζικες επιχειρήσεις να συμμετέχουν στις διεθνείς προμήθειες στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να προστατεύσουμε και την ιδιοκτησία της τεχνολογίας. Ε, πιστεύω ότι στο μέλλον η κατεύθυνση προς τα οποία θα πρέπει να κινηθούμε είναι το win-win, να έχουμε μια ομοιβαία υποφελή σχέση με την Κίνα. Ευχαριστούμε, ο εκπρόσωπος των σοσιαλιστών δεν παρευρίσκεται, αλλά η Μακολάδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την ανακοίνωση και για το έγγραφο το οποίο είναι πλήρως ε, πιστεύω και καλύπτει όλα τα σημεία που πρέπει να καλυφθούν. Ωστόσο αυτό που είναι απογοητευτικό είναι το σύνηθες. Η ανακοίνωση ε, του Συμβουλίου τόσο αποδυναμωμένη που είναι πλέον. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η θέση των διαφόρων κρατών μελών στο Συμβούλιο ώστε να πλησιάσει, να προσεγγίσει στη θέση που κεφράζεται μέσω της ανακοίνωσης. Επίσης, μας είπατε ότι η αφήγηση έχει ξεκινήσει ως προς την Κίνα, υπογραμμίζοντας δηλαδή τις απειλές ενάντια των προκλήσεων, αλλά ίσως δεν είναι αυτή η γλώσσα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαιότητα, εγώ θα έλεγα. Είναι σημαντικό να κάνουμε μια μετάβαση σε ένα πλαίσιο σχέσεων που να βασίζονται στο διάλογο. Όπως έλεγε και ο πρόεδρος Σάφετ, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις, αλλά και συνολικά τις σχέσεις μας και να είναι αμοιβαίε αυτές. Η Κίνα ήταν υπερβολικά μακριά από τη θέση μας στα μέτρα που χρησιμοποιούσε στο διεθνές εμπόριο, γιατί το επιτρέψαμε. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μέτρα που θα εξασφαλίζουν αυτή την αμοιβιότητα. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι η Κίνα θα πρέπει να συμμορφωθεί, να αποδεχθεί τους διεθνείς κανόνες του ΠΟΕ. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς αξιολογείται τη θέση της Κίνας σχετικά με την πολυμέρεια, την μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. και τι θα συνέβαινε εάν δεν ευρισκόταν καθόλου η Κίνα σε αυτό το πλαίσιο έστω της θεωρητικής δέσμευσης. Επίσης σχετικά με αυτό που είπατε πριν για το διεθνές μέσο των δημοσίων προμηθειών, νομίζω ότι αυτό είναι το εκρεμές στοιχείο ως προς τη νέα πολιτική εμπορικής αμήνης. Γνωρίζω τη θέση της Κομισιόν. Αυτή αποτυπώνεται στην ανακοίνωση, αλλά θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία από το Συμβούλιο για τις πραγματικές δυνατότητες που θα έχουμε, ώστε να αναπτύξουμε το μέσο αυτό. Και τέλος, έχω την εντύπωση ότι η Κίνα αναπτύσσει με μεγάλη αποτελεσματικότητα την οικονομική της στρατηγική, τακτική και ήθελα να καταλάβω τι μέσα έχουμε εμείς στην Κίνα για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας. Μέσω των κρατών μελών που πάντα είναι δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει πώς μπορούμε να ασκήσουμε μια ενιαία κοινή διπλωματική προσπάθεια, διπλωματία σχετικά με επενδυτικές κινήσεις και τα υπόλοιπα που γίνονται για τα επιμέρους πρωτόκολλα, για τα κράτη-μέλη, για το δρόμο του μεταξιού κτλ. Η ΣΥΑΡ, ποιος θα λάβει το λόγο. Θα μιλήσω εγώ, Πρόεδρε εκ μέρου τη ε, κυρία Μακλάρκιν. Συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να είμαστε αφελεί. Η Κίνα θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να επιτύχει τι δέσμευσει που έχει αναλάβει για την ε, ε, υποχρεωτική μεταφορά τεχνολογία. Πρέπει να εφαρμόσει τι αρχέ και το πνεύμα τη συμφωνία του και των κανόνων του ΠΟΕ. Αλλά οι λύσει των προβλημάτων τη κινέζικη οικονομία δεν μπορεί να είναι ο περισσότερο προστατευτισμό. Μπορεί να φαίνεται άδικο να υποβάλλονται σε περιορισμούς οι εταιρείε ε, που ε, ασχολούνται με την ε, δραστηριοποίηση στην Κίνα, αλλά θα πρέπει να δούμε πώ ε, μπορούμε να ενισχύσουμε τα δυνατά μας σημεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσει τη με την Κίνα έχουν, έχουν βελτιώσει και τις, την οικονομική κατάσταση και στι δύο πλευρέ. Ναι, οι ανοιχτέ αγορέ μπορεί όντω να είναι και ευαίσθητε, ευάλωτε, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να εξετάζουμε αναπερίπτωση τι επενδύσει που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το, τον, τη συμφωνία για το screening των επενδύσεων και πρέπει να εφαρμοστεί. Το σχέδιο για το εργαλείο για τι ε, διεθνεί προμήθειε είναι πιο προβληματικό γιατί ε, περιορίζει τι αγορέ δημοσίων προμηθειών τη Ευρώπη, για τι χώρε που δεν επιτρέπουν τι ευρωπαϊκέ εταιρείε να ανοίξουν τι αγορέ του. και εδώ πραγματικά είμαστε, πρέπει να είμαστε πολύ ε, προσεκτικοί. Ε, σύμφωνα και με τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει, να, αλλάξουμε, να ανοίξουμε τι αγορέ και να έχουμε ελεύθερο εμπόριο. σω μπορεί αυτό να μειώσει τις, ε, το κέρδο και να βλάψει τι ευρωπαϊκέ εταιρείε που βασίζονται άμεσα στι υπηρεσίε ή τα αγαθά από τρίτε χώρε στα πλαίσια των διαγωνισμών που κάνουν. Η αποτελεσματική λύση δεν είναι περισσότερο λοιπόν προστατευτισμός, αλλά μια γενική μεταρρύθμιση σε επίπεδο ΠΟΕ, όπου το Πεκίνο θα υποχρεωθεί να κάνει απτή πρόοδο σε αυτά τα θέματα. Και πρέπει να συμμορφωνόμαστε βεβαίως με τους κανόνες του ΠΟΕ. Είμαστε ισχυροί για να μπορέσουμε και θα μπορέσουμε κατά πάσα πιθανότητα να επιβάλλουμε στην Κίνα να ε, συμμορφωθεί με τους διεθνείς κανόνες, αλλά πρέπει να δούμε και τον αντίκτυπο της ε, αποχώρησης της Βρετανίας από το Ηνωμένο Βασίλειο στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μια εγγύηση για ε, μια στοχοθέτηση υπέρ της ανοιχτής αγοράς και του εμπόριου. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Από το Άλντε. Όχι. Είναι κανείς. Όχι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους του σκιώδου συγητή. Ένα βασικό θέμα για μας τους φιλελευθερούς είναι η ανοιχτή, να έχουμε ανοιχτές αγορές, οι επενδύσεις φυσικά και για εμάς είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο δεν χρειάζεται να το περιπλέξουμε ακόμη περισσότερο, αλλά νομίζω ότι και με το μέσο, το οποίο έχουμε ολοκληρώσει πια, έχουμε ένα, μια δυνατότητα ολοκληρωμένη για το screening των επενδύσεων ε, στις ευρωπαϊκές αγορές. Έχουμε βρει ένα μέσο το οποίο επιτρέπει τις ανταλλαγές και το οποίο... Ε, μας δίνει μια συστηματική προσέγγιση για, τα, για τους διάφορους τομείς, έτσι ώστε την αφέλεια που μπορεί να δείξαμε στο παρελθόν να, μην, να την προλάβουμε για το μέλλον. Οπότε θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο από το ECR ε, πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ανοιχτών αγορών, αλλά να μην έχουμε και τυφλή εμπιστοσύνη βεβαίω ε, στι ανοιχτέ αγορέ. Αυτό νομίζω ότι είναι ο σωστό δρόμο και βεβαίω ε, πρέπει να αξιολογήσουμε και του κινδύνου που υπάρχουν παρόλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι θα μπορούσε ίσως να υπάρξει μεγαλύτερη οικονομική εξάρτηση και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η κοινωνική εικόνα που έχουμε ε, δεν θα την, ε, την, η κοινωνική εικόνα που υπάρχει δεν ε, θα γίνει πλέον ανεκτή. Πρέπει να δούμε τα θέματα των προσωπικών δεδομένων, της προστασίας των δεδομένων. νομίζω ότι πρέπει ξεκάθαρα μηνύματα να δώσουμε και να φροντίσουμε ώστε στο μέλλον να μην υπάρξουν και περιπτώσεις ε, κακοποίησης ή παραχάραξης αυτών των δεδομένων. Ο Χέλμουντ Σόλτς για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, Ήμουν μια μίγα στον τοίχο την ε, επόμενη εβδομάδα στη σύνοδο αυτή, γιατί πρέπει να... θα είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τι είναι το καινοτόμο εδώ, τι είναι το νέο σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια που αναφέρατε. Είχαμε μια ελαφρώς διαφορετική στρατηγική. Τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και γιατί κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση που κινούμαστε προς αυτή τη στρατηγική δηλαδή εταιρική σχέση και την στρατηγική, το στρατηγικό ανταγωνισμό στη σχέση μας με την Κίνα. Τι έχει συμβεί. Και συμφωνώ ότι ναι, πρέπει να μιλάμε με καθαρά, καθαρή φωνή και πρέπει να έχουμε υπομονή, αλλά πρέπει ξεκάθαρα να δούμε τι είναι αυτή η ανταγωνιστικ... αυτός ο ανταγωνισμός που έχουμε και πώς θέλουμε να δομήσουμε ε, αυτή την σχέση που θα έχουμε πλέον με την Κίνα. Πώς, πού θα επικεντρωθούμε στην ε, τεχνολογική ανάπτυξη, στην οικονομική ανάπτυξη, στα θέματα που αφορούν στην τεχνολογία για το μέλλον δεν μιλάω τώρα για πολιτικά ή κοινωνικά θέματα και εκεί υπάρχουν σημαντικές απαιτήσει και πρέπει να τι σκεφτούμε. Πριν από 40 χρόνια, ανεξάρτητα, είχαν, είχε πει ο πρόεδρο τη Κίνα, ανεξάρτητα από το αν η γάτα είναι άσπρη ή μαύρη, το θέμα είναι να πιάνει ποντίκια. Και αυτό οδήγησε στο ότι το 1 δις 400 εκατομμύρια πολίτες είδανε ε, να αυξάνεται η ευημερία τους και η ποιότητα ζωής τους. Ξέρουμε ότι οι Κινέζοι εδώ και πολλά χρόνια ακολουθούν αυτή την ε, γραμμή ευλαβικά. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να ζητούμε από ένα δις 400 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν όπως ζούμε εμείς. Είναι σωστό αυτό το μοντέλο ζωής. Το μοντέλο κατανάλωσης είναι σωστό για αυτούς. Τα πώς επενδύουν οι κρατικές δομές στην οικονομία. Αυτά τα θέματα πρέπει να δούμε. Αυτή είναι η συστηματική πραγματικότητα. Γιατί θεωρώ ότι είναι απολύτω αφελέ και μάλιστα είναι και λάθο να λέμε με, το δικό μα τον τρόπο θα τα πάτε καλύτερα. Εμεί θεωρήσουμε πώ θα είναι η αγορά στο μέλλον. Εμείς θα θέσουμε τα benchmark και τα πρότυπα. Όχι, είμαστε στον 21ο αιώνα. Πρέπει και εμείς να μάθουμε ότι από κοινού με άλλους ε, λαούς και με άλλες κοινωνίες πρέπει να θέσουμε τα μελλοντικά benchmarks. Εγώ συμφωνώ με όσους λένε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει βέβαια μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Βεβαίως, εκεί πρέπει να τεθούν από κοινού τα πρότυπα, να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις κτλ. Αν αυτό δεν τα καταφέρουμε, ναι, προφανώς θα υπάρξει πρόβλημα και στο οικονομικό και στο εμπορική πολιτική και στην οικονομική συνεργασία θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις. Οπότε το θέμα είναι το οικονομικό δυναμικό και της ε, λαϊκής δημοκρατίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς θα μπορέσει να ε, ε, αναπτυχθεί και εν, εν, εν ώψη της ε, Νέας Συνόδου για το μέλλον. Γιατί η κατάσταση είναι αρκετά καλή. Έχουμε μια εταιρική σχέση, μια σύμπραξη με την ε, Κίνα, μια συνεργασία. Προβληματικό είναι το να υποδεικνύουμε την στρατηγική, όπως κάνει ε, ο Τραμπ με την στρατηγική του πρώτα η Αμερική. Δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την άγουσα. Νομίζω ότι αυτό το, αυτή την πτυχή της κοινή ε, Προσέγγιση θα πρέπει να την προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζαμέ για το ΙΕΝΕΦ. E δεν έχω να πω και πολλά. Κάποιες σκέψεις μόνο. Όταν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα γεγονότα, καλό είναι τουλάχιστον να τα παρακολουθούμε. Και αυτά που ακούω σήμερα δεν με καθησυχάζουν. Γιατί συζητούμε πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση, πώς μπορούμε να αμυνθούμε, Πώς μπορεί να γίνει αυτό εάν δεν μιλούμε για προστατευτικά μέτρα, όταν γνωρίζουμε ποια είναι η οικονομική πολιτική της Κίνας. Και ακούω από ορισμένους συναδέλφους ορισμένα πράγματα που με προκαλούν προβληματισμό. Η Κίνα σήμερα φαίνεται ότι περνά μια περίοδο όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα αρχίζει να ξαναπαίρνει το πάνω χέρι και να ελέγχει τις καταστάσεις αυτό είναι μια πραγματικότητα. Επομένως, εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το τελευταίο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να παραμείνουμε αφελείς. Καν, θα είμαι σύντομος, γιατί έχω δύο γενικές παρατηρήσεις να κάνω πέρα από αυτά που ήδη ανέφεραν οι συνάδελφοι, οι οποίες έχουν σχέση με το εξής η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει την εμπορική πολιτική ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των γεωστρατηγικών αλλαγών. Και πρέπει να δούμε ποια είναι η θέση που παίρνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, όχι μόνο ανάμεσα, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και απέναντι στην Κίνα, γιατί αλλάζει η δυναμική. Επομένως, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να επιδιώξουμε μια ισορροπία. Η ισορροπία βέβαια δεν σημαίνει ότι θα εμπολίσουμε τις αρχές μας, ανάμεσα στις οποίες είναι η προσήλωση στους υφιστάμενους διεθνείς οργανισμούς, ανάμεσα τους και ο ΠΟΕ, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε και τις διάφορες ευκαιρίες οι οποίες ανοίγονται. Και αναφέρομαι εδώ πιο συγκεκριμένα στο δρόμο του μεταξιού, αυτή την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Κίνα. Ε, κάποια στοιχεία που θα έπρεπε κανείς να εξετάσει είναι τα εξής. έχουμε καλές σχέσεις με ορισμένες από τις χώρες με τις οποίες προσπαθεί να συνεργαστεί η Κίνα. Ε, και τους έχουμε δώσει, για παράδειγμα, πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και επενδυτικές ε, συμφωνίες. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε ε, τη σχέση μας με αυτές τις χώρες ως μοχλό Δεύτερον, το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαβάζω και ενημερώνω με όλο και περισσότερο για στοιχεία που έχουν σχέση με την περιοχή του Xinjiang και τον ε, τρόπο με τον οποίο η κινέζικη κυβέρνηση μεταχειρίζεται τον πληθυσμό εκεί. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και κάποια αναφορά στις ανησυχίες μας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ανακοίνωση στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής. Αυτά ήταν ουσιαστικά τα θέματα που εγώ ήθελα να θίξω. Κυρία Μινό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ο προστατευτισμός δεν πρέπει να είναι ταμπού. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας φοβίζει. Είναι κάτι το οποίο έχει διευκολύνει πολλές βιομηχανίες, πολλούς κλάδους της οικονομίας να ανθίσουν. Είναι μερικές φορές τα προστατευτικά μέτρα απαραίτητα. Θα πρέπει κανείς να αξιοποιεί ε, τα δυνατά στοιχεία της ε, οικονομίας μας, οτιδήποτε μπορεί να συνεισφέρει σε μέρες περιπτώσει στην ανάπτυξη της οικονομίας μας και την ευημερία του πληθυσμού μας. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Κίνα σε ορισμένου τομεί μας έχει ξεπεράσει. Επομένως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την αυταπάτη ότι η αγορά θα αυτορυθμιστεί και θα λύσει τα πάντα από μόνη της έχουμε δει ότι αυτή η προσέγγιση δεν οδηγεί σε βελτίωση των ε, προϊόντων ή των υπηρεσιών, ούτε βέβαια από την άλλη η επαναθνικοποίηση, η επανακρατικοποίηση επιχειρήσεων είναι πανάκια. Με λίγα λόγια, δεν θα πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι σε σχέδια τα οποία είχαμε καταρτήσει πριν από 10 χρόνια, δεδομένων των αλλαγών που έχουν γίνει. Ίσως η αποκέντρωση των υπηρεσιών να είναι μια λύση κέντρωση προς την περιφέρεια. Και το ερώτημα που θέτω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πώς θα υποστηρίξει, πώς θα βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση, αυτή την τάση. Ο κύριος Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτέλους, η Κομισιόν και η κυρία Μογκερίνη διαπίστωσαν ότι η Κίνα είναι συστημικός αντίπαλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια αυτό άλλαξε θεμελιωδώς. Στην Κίνα παρατηρούμε ένα rollback σε, μια, μια, σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς και έχει δημιουργηθεί το πιο αστυνομοκρατούμενο κράτος, το χειρότερο από τότε που υπάρχουν αστυνομοκρατούμενα κράτη. Οπότε εμείς εδώ ως Ευρωπαίοι νομίζω ότι τις αρχές μας, κυρίως τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε και πιστεύω ότι είναι καλό να μην αφαιθούμε να κάνουμε μία σύνοδο ευημερία γιατί θα μειώσουμε τη σημασία όλων αυτών των θεμάτων. Θα πρέπει να επιμείνουμε, έτσι όπως λέει και η ανακοίνωση, να δούμε απτά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε στους Κινέζους ότι αυτή τη θέση την έχουμε αποφασίσει και είμαστε ξεκάθαροι ως προς αυτό. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν οι ΙΠΑ και να κάνουμε στροφή 180 μοιρών από τη μία θέση που έλεγε παλιά συνεργασία εκεί που είναι δυνατόν και πάντα σήμερα να πούμε συνεργασία μόνο εκεί που είναι απολύτως απαραίτητη πρέπει να έχουμε μια βασική, συνεργασία, μια βασική ε, πολιτική συνεργασία. Αλλά η συνεργασία θα πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένη, με σαφεί γραμμέ. πολιτικη συνεργασια αλλιώ θα πρεπει να ειναι ξεκαθαρισμενη με σαφείς γραμμε γιατι αλλιω θα διακυβευθουν οι δικέ μα αρχέ και τα δικά μα συμφέροντα το ανοιχτό πνεύμα που ε, ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια από τον πρόεδρο, σήμερα έχει μετατραπεί σε κάτι διαφορετικό. Τότε ήθελε να ανοίξει η Κίνα προς τον ε, κόσμο και σήμερα η Κίνα κλείνει τις, πόρτες της στον ε, κόσμο και ξεκινάει απεικιοκρατικά σχέδια. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πρέπει λοιπόν εμείς πολύ συγκεκριμένα να δούμε ποια είναι τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε. ΟΠΟΕ είναι το προτιμόμενο πλαίσιο, αλλά βεβαίως διαπιστώνουμε ότι στα πλαίσια του ΠΟΕ κάποια πράγματα δεν τα λέμε. Δεν τα αναφέρουμε. Κάποιες πρακτικές στο, της ε, βιομηχανικής πολιτικής της Κίνας δεν θίγονται εντός του ΠΟΕ και η Κίνα, όταν, ε, όσο υπόσχεται, όλο υπόσχεται μεταρρυθμίσεις εμπορικές στον ΠΟΕ, και αυτό σημαίνει ότι δεν θέλει να μεταρρυθμίσει τελικά, κυρίως αν δούμε τι γίνεται με το Belt and Road. Η προσπάθεια που γίνεται εκεί είναι να αντικατασταθεί ο ΠΟΕ μέσω ενός συστήματος με κέντρο την Κίνα και να μην εξελιχθεί περαιτέρω ο ΠΟΕ. Νομίζω λοιπόν ότι και εκεί θα πρέπει πολύ συγκεκριμένα να δούμε ποια είναι τα ίδια μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εγώ είμαι κατά του προστατευτισμού, αλλά δεν πιστεύω ότι κάθε προστασία κατά του του ανταγωνισμού θεωρείται προστατευτισμός. Η διαφορά νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να προστατέψουμε χωρίς να γίνουμε προστατευτικοί. Αυτή είναι η βασική μας γραμμή, αυτή νομίζω ότι θα πρέπει να είναι η βασική μας γραμμή και θα πρέπει να, είμαστε, να επιμείνουμε και θα ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα τίμημα. Η Κομισιόν πριν λίγο καιρό, λόγω ακριβώς της κατάστασης, ε, και της ε, σύμπραξης ε, της Fusion με την Alstrom δεν την ενέκρινε και γι' αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπει στην άκρη η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τον ανταγωνισμό. Πρέπει απλώς να τροποποιηθεί και να αναλύσουμε τι γίνεται. Και κατά συνέπεια αυτός ο σούπερ γίγαντας της Κίνας έχει πλέον το πρώτο, την πρώτη του σύμβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικά να, προσε... να δούμε τι γίνεται, γιατί και για το IPI δεν πρέπει να καταντήσουμε απελπισμένοι ε, απέναντι στην Κίνα με τον τρόπο που διαπραγματευόμαστε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Και να πω και εγώ δύο λόγια. Νομίζω ότι βεβαίως πρέπει να δούμε ότι η Κίνα ως εταίρος είναι εταίρος που χρειαζόμαστε στον ΠΟΕ. Θέλουμε να υπάρχει σταθεροποίηση στον ΠΟΕ, σταθερότητα. Θέλουμε να είναι όλοι εντός του ΠΟΕ και γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς γίνεται η εξέλιξη, ο εξυγχρονισμός με θέματα για τα οποία είμαστε επικριτικοί απέναντι στην ε, Κίνα. Μιλάμε για την πνευματική διοκτησία, μιλάμε για τις κρατικές επιχειρήσεις κτλ. Αν έχουμε αυτό το στόχο, να διατηρήσουμε δηλαδή την Κίνα εντό του ΠΟΕ, πρέπει να δούμε το θέμα της εμπορική πολιτικής, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε από κοινού με την Κίνα. Νομίζω ότι με αυτή την ανακοίνωση, ναι, υπάρχει μία αλλαγή, Πίτερ, σαφή αλλαγή έναντι των θέσεων που είχαμε στο παρελθόν. Παλιά μιλούσαμε για στρατηγικό εταίρο ή ενδυνάμει εταίρο. Τώρα ξαφνικά έχουμε ένα σύστημα ανταγωνιστικό, αντίπαλο ακόμη ακόμη. Και ε, πραγματικά αυτό είναι σαφής διαφορά. Φυσικά έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό είναι σωστό και θεμητό τώρα να έχουμε κι εμείς ξεκάθαρη θέση απέναντι σε αυτή τη νέα αλλαγή. Απλώς η, η, η ισορροπία μεταξύ ξεκάθαρων λόγων και θέσεων όπως τις ε, αναλαμβάνει ο Τραμπ είναι, καταλαβαίνετε, πολύ ευαίσθητη. Εγώ δεν θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση να, πάμε, να, να ακολουθήσει την άγουσα του Τραμπ. Γιατί αυτό βεβαίως δεν θα εξυπηρετούσε και τα οικονομικά μας συμφέροντα. Πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη θέση απέναντι στην ε, Κίνα χωρίς όμως να διακυβεύσουμε τις δικές μας αρχές και αξίες. Νομίζω αυτός είναι ο πυρήνας των δραστηριοτήτων μας από εδώ και μπρο. Τώρα η προσπάθεια του, της απομόνωσης ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι κομμάτι των α, δικών μας δραστηριοτήτων. Πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε αυτά τα 10 μέτρα τα οποία λίγο πολύ είναι ρεαλιστικά για το εγγύ μέλλον, αλλά ίσω θα πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο πιο μακριά, πιο στρατηγικά για το απότερο μέλλον. Αυτό είναι ένα σημείο που μπορούμε νομίζω να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά και το ερώτημα του πώς πάμε παραπέρα είναι σημαντικό. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη. Νομίζω ότι αυτό είναι απλώς το ξεκίνημα μιας συζήτησης που θα συνεχιστεί στα επόμενα δύο χρόνια. Σήμερα ακούσαμε πολλές πτυχές αυτής της περίπλοκης σχέσης ε, αποπειραθήκαμε εδώ μέσω μιας ανακοίνωσης να συμβάλλουμε στην συζήτηση του Συμβουλίου και με την ευκαιρία εξετάσαμε το σύνολο της σχέσης μας με την Κίνα με τρεις βασικούς στόχους. Εμβάθυνση των δεσμεύσεων για να έχουμε κοινά συμφέροντα διεθνώς, μια πιο ισόρροπη και ισοσταθμισμένη σχέση και τρίτον να προσαρμόσουμε τις δικές μας εμπορικές και οικονομικές πολιτικές προς την πραγματικότητα. Υπάρχει η αναγνώριση ότι ο ρόλος της Κίνας έχει αλλάξει. Δεν είναι πλέον μια αναπτυσσόμενη χώρα, λέει ο Η Κίνα είναι ένας παγκόσμιος παίκτη και πολύ σημαντικός. Και είναι και ηγέτιδα τεχνολογικά. Είναι ένας ε, στενός εταίρος με τον οποίο διαπραγματευόμαστε. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Είναι οικονομικός ανταγωνιστής, είναι συστημικός ανταγωνιστής και αντίπαλος με εναλλακτικά πρότυπα διακυβέρνησης και μας ανταγωνίζεται και στις αγορές, τις τρίτες αγορές εξαγωγών. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και το είχαμε συζητήσει και με τα κράτη-μέλη στην Κορεπέρ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ενωμένη απέναντι στην Κίνα. Εδώ πρέπει να ξεπεράσουμε λοιπόν κάποιες στενές εθνικές προσεγγίσεις για τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχουμε για την Κίνα. Είναι κρίσιμη σημασία. και συνολικά για τις ενωσιακές σχέσεις με την Κίνα και για τις εθνικές όμως επιμέρους σχέσεις. Για παράδειγμα σε αυτό το διεθνές μέσο για τις ε, προμήθειες. Εδώ πρέπει να φτάσουμε σε ισότιμους κανόνες παιχνιδιού κάποιος από τα μέλη αναφέρθηκε στην αμοιβαιότητα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία πρόσβαση στην αγορά προμηθείων της Κίνας. Δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια προσχώρησης στο, στην κοινή συμφωνία για τις προμήθειες, για τις δημόσιες προμήθειες. Εμείς προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε τη σχέση αυτή, να δώσουμε κίνητρα στην Κίνα να ανοίξει την αγορά της των προμηθειών. Εδώ ποια είναι η πρόκληση. Έχουμε μια χώρα τεράστια σε μέγεθος και σε οικονομικό μέγεθος και σε πληθυσμιακό μέγεθος και ακολουθεί ένα διαφορετικό μοντέλο από το δικό μας, τον κρατικό καπιταλισμό. Και εδώ θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ε- κρατικών ενισχύσεων, των κρατικών επιδοτήσεων για το οποίο δεν έχουμε κανόνες στον ΠΟΕ. Όπου είναι το κατάλληλο βήμα, αλλά πρέπει να επικαιροποιηθούν οι κανόνε του ΠΟΕ, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Εργαζόμαστε με την Κίνα διμερό για τα θέματα τη μετερρύθμιση του ΠΟΕ, συνεργαζόμαστε με την Ιαπωνία, με τι ε, ΗΠΑ. Πρέπει να δούμε λοιπόν την υφιστάμενη σχέση στα πλαίσια των διαφορών και των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. οι Αμερικανοί έχουν υποβάλει κάποια διάγνωση και πρέπει να δούμε αν την συμμεριζόμαστε και βεβαίως να έχουμε και τα μέσα για να ακολουθήσουμε μια αντίστοιχη κατεύθυνση με την Αμερικανική. Οποιαδήποτε πάντως συμφωνία προκύψει από τις διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΠΟΕ και να επιβάλλεται σε πλαίσιο πολυμέρειας. Όλα αυτά θα δραματίσουν ρόλο στην δήλωση της Συνόδου, όπως φαντάζεστε. Και εδώ αυτό είναι ένα θέμα επί του οποίου δίνουμε ακόμα μάχη για την ακριβή διατύπωση, ορολογία, με τους Κινέζους ομολόγους. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη συμφωνία για την κοινή δήλωση. Υπάρχουν κρεμοί ανοιχτά ζητήματα αυτή τη στιγμή που μιλούμε. και θα πρέπει να επανέλθω σε αυτό στην επόμενη αναφορά που θα σας κάνω για την σύνοδο. Ευχαριστούμε Πίτερ λέει ο Πρόεδρος. Ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτό είναι η πιο αμυντική όψη του νομίσματος ως προς την Κίνα. Ίσως να μας λείπει η επιθετική όψη. Δηλαδή να δούμε τις εσωτερικές μας δομές που δεν είναι αρμοδιότητα της δελτα αλλά και ως προς την νομοθεσία τη διατάξη του ανταγωνισμού της δικές μας. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξυγχρονίσουμε την εσωτερική μας πολιτική υπό το φως αυτής της διεθνούς κατάστασης. Αυτό πιστεύω εγώ. Ευχαριστώ όλους. Και με αυτό κλείνουμε το σημείο 13 και πάω απευθείας στο σημείο 14 το οποίο συνήθως έπεται του 13. Εδώ έχουμε την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις άμεσες εξωτερικές ενισχύσεις τρίτων χωρών δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που άπτεται και του προηγούμενου και θα δώσω τον λόγο στον κύριο Κάρλο Πετινάτο, επικεφαλής της ομάδος της υπηρεσίας για την πολιτική επενδύσεων από τη ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν ο Πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε στο State of the Union ότι η Κομισιόν θα πρότεινε ερευνητικούς ελέγχους screening για να συνεννοούμεθα. Θα πρότεινε επίσης μια ομάδα συντονισμού με τα κρατη για το FDI screening και μια ενδελεχή έκθεση για τις εξελίξεις στα θέματα των επενδύσεων τρίτων χωρών, για τα θέματα γεωγραφικών ενδείξεων, προέλευσης, ιδιοκτησίας λοιπά. Εξού και δημοσιεύσαμε την έκθεση 13 Μαρτίου μετά την ανάληψη της δεσμεύσεως. Οι δύο λόγια για τους οποίους θέλαμε να δούμε λίγο τις διεθνείς τάσεις, τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές, το πώς έχουν τα πράγματα, δεν ήταν μόνο για να δούμε τα επίσημα μεγέθη και τις στατιστικές, αλλά για να πάμε πέραν αυτού και να δούμε ποιος βρίσκεται πραγματικά πίσω από τις επενδύσεις που γίνονται στην Ευρώπη. Και συχνά ο πραγματικός δικαιούχος, ιδιοκτήτης, δεν είναι αυτός που εμφανίζεται στα επίσημα έγγραφα. Έπρεπε λοιπόν να αναπτύξουμε μια νέα τράπεζα δεδομένων επί τη βάση εμπορικά διαθέσιμων στοιχείων, orb, έφη, αυτά τα συνδυάσαμε για να δούμε τους τελικούς δικαιούχους. Συστήσαμε λοιπόν μια νέα τράπεζα δεδομένων, την, την τράπεζα δεδομένων για τους ε, επενδύσεις τρίτων χώρων. Τα πορίσματα. Πρώτα απ' όλα το βλέπετε αυτό και στην ε, σύνοψη, την περίληψη της έκθεσης. Υπάρχουν διάφορες άλλες λεπτομερείς ε, πληροφορίες και στοιχεία, αλλά θα επικεντρωθώ στα πιο σημαντικά. Για να έχετε μία εικόνα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τι σημαίνει επιχειρήσεις με ξένους ιδιοκτήτες αυτό το γράφημα είναι λίγο δύσκολο ίσως να αντιληφθεί κανείς τι σημαίνει. Στην έκθεση είναι πιο εύκολο. Στα αριστερά βλέπετε τον αριθμό των επιχειρήσεων εξαρτητούς μεγέθους. Πόσες επιχειρήσεις έχουν ξένους δικαιούχους ιδιοκτήτες στην Ευρώπη. Στο μπλε είναι οι εισηγμένες. Συνήθως μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οι κόκκινες είναι ιδιωτικές. Γνωρίζουμε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία εν πολλής αποτελείται από μη εισηγμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες. Και αν η συνολική, το συνολικό ποσοστό των ξένων δικαιούχων είναι 3% για τις ιδιωτικές, είναι πολύ ψηλότερο 5 με 9% για τις εισηγμένες. Και αυτές είναι μεγαλύτερες όπως σας έλεγα. Μεγαλύτερες σημαίνει υψηλότερης καινοτομίας, υψηλότερης παραγωγικότητας. Στα δεξιά βλέπει κανείς ακόμη πιο εντυπωσιακά σε πλαίσιο περιουσιακών στοιχείων γιατί ακόμα και αν ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι 9% των εισηγμένων, στα περιουσιακά του στοιχεία η συμμετοχή είναι πολύ μεγαλύτερη. Το, φτάνει το 45% των εισηγμένων στην Ευρώπη και το 32% των ιδιωτικών. Δηλαδή, ξένοι επενδυτές έχουν σημαντικό μερίδιο σε μεγάλες εταιρείες, μεγάλες επιχειρήσεις. Εδώ Βλέπετε τους ε, ξένους δικαιούχους και επενδυτές και πόσο σημαντική είναι σε συγκεκριμένους τομείς κλειδιά της οικονομίας. Πετρελαιοειδή, φαρμακευτικά, ηλεκτρονικά, ορυκτά, ασφάλειες, για παράδειγμα, είναι οι πιο σημαντικοί τομείς. Όπου οι ξένοι επενδυτές φτάνουν και το 65% στα πετρελαιοειδεία ή άνω του 50 στα φαρμακευτικά. Για τις πηγές τώρα προέλευσης, ποιοι είναι αυτοί οι επενδυτές. Παραδοσιακά βεβαίως ηγούνται και επικυριαρχούν και ακόμα είναι η αλήθεια αυτό οι βορειοαμερικανοί επενδυτές μετά οι χώρες 7 Ελβετία, Νορβηγία όλοι οι άλλοι είναι ακόμα ε, σχετικά μικροί ως προς τα, τη συμμετοχή σε περιουσιακά στοιχεία όμως ως προς τις νέες συμφωνίες και νέες συγχωνεύσεις η τάση αλλάζει σημαντικά. Εδώ η ανάδυση της Κίνας μόλις, μόλις που φαίνεται στο συνολικό μερίδιο περιουσιακών στοιχείων είναι 3%, είναι, δεν μπορείτε καν να το δείτε, σχετικά με 6% που είναι μόνο Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από την ε, Κίνα, ή 11% για τις χώρες ΕΦΤΑ, ή 60% για Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Όμως η εικόνα μπορεί να ερμηνευτεί και διαφορετικά. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπουμε την αυξανόμενη ποικιλία προέλευσης των ξένων επιχειρήσεων και των ξένων δικαιούχων. Εδώ δεν μιλούμε για περιουσιακά στοιχεία, μιλούμε για επιχειρήσεις. Οι παραδοσιακοί επενδυτές, συγκρίνοντας την καφέ με την γκρι στήλη, όπου κατέρχεται το μερίδιο των ΗΠΑ, ποιος έχει αυξήσει πολύ, είναι η Κίνα και άλλα μέρη του κόσμου. Είναι ο αριθμό δηλαδή των επιχειρήσεων των αναδυόμενων αυτών οικονομιών, και αυτό είναι η κόκκινη γραμμή, που έχει αυξηθεί πολύ. Ρωσία, Κίνα, Ινδία και άλλα μέρη του κόσμου έχουν αυξηθεί σημαντικά. Εδώ τώρα μιλούμε για εξαγορές. Όπου και πάλι η τάση δείχνει ότι οι νέοι συμμετέχοντες, οι νέοι παίκτες, οι αναδυόμενες οικονομίες είναι πολύ πιο σημαντική παρά τη συνολική του συμμετοχή. Ε, εξακολουθεί Αμερική, Καναδά, ΣΕΦΤΑ να είναι οι μεγαλύτεροι εξαγοραστές. Αναπτυσσόμενη Ασία, η Ιαπωνία, Κορέα, Σιγκαπούρη λέει ο μιλητής. Εξαιρετικά υψηλά στο 9 και κάτι offshore χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κέντρα, θα επανέλθω, άνω του 8%, offshore, αυτή είναι η πηγή, Κίνα 6,5% των εξαγορών. Που σημαίνει ότι οι εξαγορές είναι πολύ πιο σημαντικές από το συνολικό τους μερίδιο στα περιουσιακά στοιχεία και αν δούμε τους τομείς οι παραδοσιακοί επενδυτέ, οι ΗΠΑ, ΕΦΤΑ, εμφανίζονται σε όλα τα πεδία και με υψηλότατο επίπεδο διαφοροποίησης σε όλο το φάσμα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αναπτυγμένη αστεία Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, πιο εστιασμένη. νέοι άλλοι επενδυτές γίνονται όλο και πιο εμφανείς σε διάφορους τομείς με υψηλότατο βαθμό εξειδίκευση. Εδώ μιλούμε για τα offshore, για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Κίνα στην ε, κατασκευή αεροσκαφών εξειδικευμένα μηχανήματα, Ινδία στα φαρμακευτικά κτλ. Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες στην έκθεση. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι οι αναδυόμενοι παίκτες είναι πιο εξειδικευμένοι. Κοιτώντα τώρα το είδο των επενδύσεων, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το διαβάσει κανεί ίσω, αλλά θα σα το εξηγήσω. Έχουμε τα χαρακτηριστικά του κάθε επενδυτή, του κάθε αγοραστή. Συνήθως μιλούμε για βιομηχανικές ε, επιχειρήσεις, το οποίο δεν δείχνεται καν σε αυτό το γράφημα, είναι πολύ πιο ψηλά δηλαδή από αυτά. Τα υπόλοιπα λοιπόν πλην βιομηχανικών είναι το μερίδιο των χρηματοπιστωτικών και τραπεζών και ασφαλιών που είναι η πράσινη γραμμή έχει κατέλθει σημαντικά σε σχέση με άλλους παίκτες όπως είναι investment funds επενδυτικά ταμεία ιδιωτικά ανεξάρτητοι ιδιώτες και κρατικοί φορείς και εδώ εννοούμε τα ίδια τα κράτη και όχι κρατικές επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν και αυτές να είναι βιομηχανικές. Νέο είδος, νέα είδη λοιπόν επενδυτών. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη τάση μετατροπής του οικονομικού πλαισίου σε χρηματοπιστωτικούς τίτλους. και κοιτώντας την πηγή, την προέλευση των αγοραστών, εδώ έχουμε ισχυρή παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κέιμαν και της Ελβετίας. Αλλά υπάρχει πολύ σημαντική αύξηση ιδιωτών ή οικογενειακών ταμείων από το 31 στο 197 λέει ο μιλητής. Εδώ μιλούμε για κυρίως Ελβετούς, Αμερικανούς, Ρώσους, Νορβηγούς. Κατόχους διαπατηρίων δηλαδή. Αν δούμε τις κινέζικες τώρα επενδύσεις ανά είδος, χωρίς να κοιτούμε τα απόλυτα μεγέθη, ξεκίνησαν αργά τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι κρατικές κινέζικες επιχειρήσεις που είναι το μπλε, πάντοτε ήταν υψηλότερες από τις ιδιωτικές, εκτός του έτους 16, που ήταν έτος έκρηξης εξαγορών για την Κίνα. το οποίο αποτυπώνει και το χαρακτήρα της οικονομίας στην Κίνα και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή. Αυτό εδώ είναι η τελευταία διαφάνεια. Την, το μερίδιο στην απασχόληση. Περί το 17% των απασχολουμένων συμπεριλαμβάνεται στην τράπεζα αυτή δεδομένων, δηλαδή από επιχειρήσεις των οποίων οι δικαιούχοι είναι ξένοι υπήκοοι. Αυτά είναι τα πορίσματα κλειδιά στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Thanks Σας ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις. Helmut, κύριε Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε και αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θα έλεγα ότι είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε μια ξεκάθαρη τάση ενίσχυσης της Κίνας και άλλων ανδυόμενων οικονομιών. Άρα παρόλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι κατά κύριο λόγο οι ξένες επενδύσεις προέρχονται από τους παραδοσιακούς ε, και χώρες επενδυτές. Και επίσης παρατηρούμε ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό των offshore, 11%. σε αριθμό επιχειρήσεων και 4% σε στοιχεία ενεργητικού. Σε όλη την Ένωση φυσικά. Δεν ήταν και τόσο καθαρό, αλλά θα έλεγα ότι τα στοιχεία φαίνεται να καταδεικνύουν ότι αυτή η τάση είναι αυξητική το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα της φορολογίας, της ε, φοροαποφυγής και του ξεπλήματος μαύρο χρήματο για τους σκοπούς για τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιούνται αυτές οι offshore. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι προς την Επιτροπή πώς εσείς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτή τη αυξανόμενο ποσοστό ξένων επενδύσεων που προέρχονται από φορολογικούς παραδείσους. Κάτι ακόμα είναι ότι διαπιστώνουμε να υπάρχουν όλο και περισσότερες εξαγορές από εξωτερικούς επενδυτές, ε, αυτό που είπατε πριν, ότι μετατρέπεται η οικονομία σε όλο και περισσότερο σε χρηματοπιστωτικούς τίτλους. Το οποίο σημαίνει όμως ότι εκτιθέμεθα όλο και περισσότερο στην κερδοσκοπία και στις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών. Πώς μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει αυτό και πώς μπορεί να ενισχύσει α, πώς, τι, πώς έχουμε αξιολογήσει, τι σημαίνει αυτό για την πραγματική οικονομία. Επίσης, το, ο νέος μηχανισμός screening ε, εξετάζει και αυτό το ζήτημα, δηλαδή τον κίνδυνο που δημιουργεί το γεγονός ότι έχουμε ξένες απενδύσεις όχι μόνο από τις αναδυόμενες νέε οικονομίες, αλλά επίσης από αυτού τους φορολογικούς παραδείσους και τις offshore. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι μάλλον η τελευταία φορά που θα πάρω το λόγο εδώ, επομένως θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τον πρόεδρο και επίσης και τον προκάτοχό του, τον ε, καθηγητή Μαρέρα. Πολλοί θα τον θυμούνται. Αυτό που ακούσαμε νομίζω, είναι μια πολύ ξεκάθαρη παρουσίαση των ε, στοιχείων, των πραγματικών στοιχείων για τις ξένες επενδύσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και νομίζω το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ήταν το τελευταίο, δηλαδή 17% των απασχολούμενων στα 28 κράτη-μέλη της Ένωσης εργάζονται για κάποιες ε, επιχειρήσεις οι οποίες ε, ανήκουν σε ξένους υπηκόους, το οποίο μου φαίνεται τεράστιο. Αυτό που δεν άκουσα και εξού και η ερώτησή μου είναι το εξή. Διαβάζω εδώ από ένα δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέει, παρά το ε, μια, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανοιχτή προς ξένες επενδύσεις όμως αυτές οι επενδύσει θα πρέπει να παρακολουθούνται έτσι ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο τα στρατηγικά ε, συμφέροντα της Ένωσης και ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο ε, κανονισμό ο οποίος μας προστατεύει ευαίσθητους τομείς της οικονομίας όπως για παράδειγμα η αεροναυπηγική, το διάστημα, η ενέργεια κτλ. Ε, ο κύριος Φρανκ Προύστ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρω ότι δεν εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχω διαπιστώσει ότι πολλέ συχνά οι απόψει του ταυτίζονται με αυτέ τι επιτροπέ. Τις επιτροπές. Λέει ότι αυτή η παρακολούθηση των δημοσίων, ξένων δημοσίων επενδύσεων θα πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Το οποίο σημαίνει ότι η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει μια πολύ πιο διαφορετική προσέγγιση από αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Γαλλία έχει επιλέξει κάποιου στρατηγικού τομεί και απαγορεύει ξένες επενδύσεις στον τομέα αυτών. Για παράδειγμα, ε, για εκείνους, για, για τους Γάλλους, αντιλαμβάνονται τον τομέα της διατροφής ω ε, ως στρατηγικό τομέα. Είναι άλλη η στρατηγική τομή για την, το Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ δεν προσπαθώ να κάνω αξιολογικές κρίσεις, απλώς αναφέρω τι συμβαίνει. Έχουμε μια πολύ πιο ανοιχτή οικονομία εμείς. Για παράδειγμα, επιλέξαμε, επιτρέψαμε στην EDF Electricité de France να επενδύσει στο ενεργειακό μας δίκτυο. Και έρχομαι στο ερώτημά μου. Μας παρουσιάσατε τα στοιχεία. Το, στο πλαίσιο όμως το οποίο βρισκόμαστε, αντιλαμβανόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρμοδιότητες οι οποίες της επιτρέπουν όχι μόνο να παρακολουθεί, αλλά επίσης και να επηρεάζει ή ακόμα και να προλαμβάνει τις ξένες επενδύσεις στο βαθμό που μπορείτε να μας τα ανακοινώσετε αυτά. Πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει τις αρμοδιότητες της στη βάση αυτών των στοιχείων που συλλέξατε. Ευχαριστώ. Ίνμα. Ευχαριστώ. Να πω πρώτα απ' όλα ότι μου φάνηκε πληρέστατη η παρουσίαση και ευχαριστώ τον εκπρόσωπο Έχετε μία ανάλυση αναχώρα, ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, ποιο είναι το μερίδιο αναχώρα και αναείδος επένδυσης. Και αν δεν έχετε αυτές τις πληροφορίες, έχετε την πρόθεση να τις αναπτύξετε, να τις καταγράψετε. Για τις ερωτήσεις του κυρίου Σόλτς ε, μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε πώς θα έχει η στρατηγική σχετικά με επενδύσει που προέρχονται από φορολογικού παραδείσους ή πηγαίνουν προς φορολογικού παραδείσους και για το κατά πόσον ε, είναι ε, δίκαιο και σωστό για τους κανόνες ανταγωνισμού να έχουμε φορολογικούς παραδείσους και εντός Ευρωϊκής ε, Ένωσης. Τώρα για την στρατηγική της Κίνας και για τον δρόμο του μεταξιού. Η υπογραφή πρωτοκόλων με την Κίνα από συγκεκριμένα κράτη-μέλη σε αυτή την κατεύθυνση ε, πώς συνδυάζεται με το μηχανισμό screening στον οποίο αναφερθήκατε για στρατηγικούς τομείς. Το κάθε κράτος μέλος βεβαίως έχει την κυρίαρχη δυνατότητα να κινηθεί όπως πιστεύει, αλλά ε, είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενες ευκαιρίες στο Συμβούλιο το θέμα αυτό του στρατηγικού μηχανισμού, δηλαδή πώς θα δεσμευθούν τα κράτη-μέλη προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Όπως είπε ο συνάδελφος, πολλοί όντως ε, απασχολήθηκαν μέσω των ε, εξωτερικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικό μου το ερώτημα είναι, έχετε κάποια ξεκάθαρη, κάποιο όραμα και εικόνα ξεκάθαρη για την ε, συμπεριφορά των επενδύσεων προς, προς το εργατικό δυναμικό. Έχω, ας πούμε, μία περίπτωση εγώ στη δική μου την εκλογική περιφέρεια, όπου μία μεγάλη αυτοκίνητο βιομηχανία που έχει μάλιστα και πολύ, καλό, πολύ καλή θέση σύμφωνα με τη Standard Poor's Έχουν επενδύσει σε διάφορες ε, χώρες, οι συνθήκες βεβαίως είναι διαφορετικές στις άλλες χώρες και χρησιμοποιούν την θέση τους μέσω των επενδύσεων στο να πιέζουν τους εργαζομένους. Είναι μοναδική η περίπτωση αυτή. Έχετε εσείς ε, κάποιο προοπτική πιο καθαρή ή κάποια διαφορετική άποψη από το πώς φέρονται οι επιχειρήσεις μέσω των λόγων μάλλον των εξωτερικών επενδύσεων στο εργατικό δυναμικό. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και πολύ σημαντικές. Η παρουσία των ε, κέντρων offshore, των οικονομικών κέντρων offshore ως πηγή αυξάνεται. Οι λόγοι νομίζω είναι σαφείς. Μιλήσατε κι εσείς. Κυρίως για, φορο, για λόγους φοροαπαλλαγής, για βελτιστοποίηση των φορολογικών εσόδων, ή για άλλους ε, λόγους. Γεγονός πάντως είναι ότι είναι όλο και πιο σημαντική αυτή η πόρη και αν έχετε χρόνο δείτε ένα πεδίο στη σελίδα 12 της έκθεσης που μελετά για το ποιος επενδύει στους, ε, στους οικονομικούς, στα οικονομικά κέντρα offshore. Ξέρουμε δηλαδή ότι υπάρχουν ε, κάποιες ε, πηγές, αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι πίσω τους. Ξέρουμε όμως ποιος επενδύει σε αυτές αρχικά. Και είναι αρκετά αξιόπιστο περίεργο το πώς οι Αμερικανοί επενδυτές ε, ε, βασίζονται κυρίως σε συγκεκριμένα κέντρα, όπως οι Βερμούδες ας πούμε, ενώ οι Κινέζοι ενδιαφέρονται για άλλα κέντρα, όπως ας πούμε τα, οι Βρετανικές Παρθένες νήσι. 80% οι επενδύσεις εκεί είναι από την Κίνα. Οπότε μπορείτε έτσι γενικώ να έχετε μια εικόνα του ποιο βρίσκεται από πίσω. Βεβαίω υπάρχουν και πολλοί Ευρωπαίοι που επενδύουν και μετά επανεπενδύουν. To uh, uh, Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να επιβάλλουμε φόρους που θα είναι πληρωτέοι και στην οικία χώρα. Είπαμε ότι αυτό, αυτή η έκθεση θα ε, πήγαινε και θα συμπληρώνε και το ε, screening του FDI. Προ το παρόν προσπαθούμε να δούμε τα θέματα ασφάλειας. Δεν μιλούμε για θέματα απαλλαγή. Οπότε δεν έχω πραγματικά την αρμοδιότητα να το μελετήσω εγώ αυτό, αλλά θέλαμε για λόγους ασφάλειας να καταγράψουμε και αυτά τα στοιχεία, την ε, προέλευση δηλαδή. Αυτό ίσως να είναι αρκετά ενδιαφέρον για το μέλλον, για την περίοδο της εφαρμογής. Αλλά αυτό είναι ο μόνος λόγος, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το θέμα της ασφάλειας. Τώρα, πώς απαντούμε στο, στον ξενόμενο αριθμό αυτών των κέντρων και τα διάφορα, τα διάφορα ταμεία που αναδύονται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα στη σημερινή οικονομία. Ένα μεγάλο κομμάτι του κεφαλαίου που είναι διαθέσιμο πηγαίνει μέσω αυτών των μέσων σε επενδύσεις. Αλλά επειδή δεν είναι κατασκευαστικές εταιρείε που επενδύουν, δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη είναι ασταθείς. Μιλούμε για ε, ξένες επενδύσεις, δηλαδή χρήματα που μπαίνουν σε ε, μακροπρόθεσμους, ε, μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Δεν μιλούμε για χαρτοφυλάκια και σχετικές επενδύσεις. Είναι κάτι άλλο αυτό τελείως. Μιλούμε για φυσικούς, ε, φυσικά περιουσιακά στοιχεία εδώ. Δεν υπάρχει λοιπόν ιδιαίτερη απόδειξη πτυτικότητας εδώ ή αλλαγών. στην ιδιοκτησία της επένδυσης. Και σε κάθε περίπτωση πάλι το θέμα αυτό δεν ήταν στο πεδίο εφαρμογής της ε, έκθεσης, να δούμε δηλαδή τη συμπεριφορά. Τώρα, τι θα πει αυτό για την πραγματική οικονομία. Νομίζω ότι θα πει ότι η σημερινή οικονομία έχει ως εξής. Πολλά από αυτά τα μέσα, ε, στα εξωτικά ταμεία, ας πούμε, από τον Καναδά, είναι πάρα πολύ σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα. Εξασφαλίζουν ότι πολλές από τις εταιρείες μας μπορούν να λειτουργήσουν και διαδημιουργούνται και θέσεις εργασίας. Δεν είναι δηλαδή πάντα ανησυχητική η τάση, έτσι είναι η πραγματικότητα. Έτσι κινείται το κεφάλαιο, έτσι χρησιμοποιείται το κεφάλαιο παγκοσμίω. Είπα ότι ο στόχος του screening είναι αυτός που είναι. Είπαμε ποιο είναι το πλαίσιο που έχουμε δημιουργήσει. Ο στόχος δεν είναι να δούμε την, ε, το αν υπάρχει κερδοσκοπία ή όχι μιλούμε για άμεσες ξένες επενδύσεις, που είναι, που είναι θέμα κυρίως ελέγχου και είναι μακροπρόθεσμες, οπότε δεν γίνεται να έχουμε πολύ εύκολα ε, κερδοσκοπία, αλλά ο στόχος είναι να δούμε τους, ε, τον κίνδυνο ασφάλειας που μπορεί να υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ φτάνουμε στο κατά πόσο η Ευρώπη που προστατεύει και το κατά πόσο αυτή η φράση σημαίνει ότι θα αλλάξουμε και στρατηγική ή αν θα αντικαταστήσουμε τα κράτη-μέλη, τις αρχές των κρατών μελών. Όχι, το είπα πολλές φορές. Το πλαίσιο εγγυάται συνθήκες συγκεκριμένες και διαδικαστικές απαιτήσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για όλους τους εθνικούς μηχανισμούς screening. Και βεβαίως χρειάζεται και συνεργασία για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και η Κομισιόν, όπως ξέρετε, θα, εκφράζει, θα ε, εκδίδει τις ε, γνωμοδοτήσεις τις ε, συστάσεις για μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων. Δεν υπάρχει δυνατότητα κυρίας, δεν υπάρχει δυνατότητα βέτο, αλλά μπορούμε να καταγράψουμε καταρχάς τους κινδύνους ασφαλείας και ίσως να κάνουμε και κάποια συστάσεις για μέτρα μετριασμού. Σε περιπτώσεις τώρα που ε, η Κομισιόν μπορεί να δράσει, βέβαια δεν μπορώ να σας πω ποια είναι τα σχέδια της Κομισιόν, γιατί η Κομισιόν δεν έχει σχέδια να ε, κινηθεί προς μία ή την άλλη κατεύθυνση σε αυτό το πεδίο. Θέλουμε να κάνουμε κάτι που δεν ε, έχει ξαναγίνει στην Ευρώπη, δηλαδή να δούμε ποιο επενδύει, να μάθουμε ποιος επενδύει και να μοιραστούμε αυτέ τι πληροφορίε ώστε να καταγράψουμε τον κίνδυνο αν υπάρχει. Γιατί σήμερα αυτό δεν συμβαίνει. Γίνεται σε κάποια κράτη-μέλη ε, μεμονωμένα, αλλά δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ κρατών μελών ή μεταξύ του κράτου μέλου και τη Κομισιόν που μπορεί όντω να επηρεάζονται από θέμα ασφάλεια. Ε, από επενδυτέ που επενδύουν σε ένα γειτονικό κράτο. Αυτό σήμερα δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Και μέσω του κανονισμού FDI θα μπορέσουμε να καταγράφουμε καταρχά ποιοι είναι οι κίνδυνοι και να δούμε αν υπάρχουν μέτρα μετριαστικά. Τώρα, για τα κατακαιρματισμένα δεδομένα. Ναι, δεν ήταν ο στόχος μας, προφανώς. Εδώ έχουμε μία δομή που βασίζεται σε βάσεις δεδομένων με εκατοντάδες χιλιάδες στοιχεία για εταιρείες. Ήτανε μια αρχιτεκτονική που έπρεπε να δημιουργηθεί για να γίνει αυτή η βάση δεδομένων. Μπορεί να γίνει βέβαια για να βρει κανεί που βρίσκονται, αλλά σήμερα δεν το έχουμε κάνει, δεν έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά. Στο μέλλον όμω είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε. Να δούμε δηλαδή ένα κράτο μέλο στα στοιχεία. Τώρα για του ε, φορολογικού παραδείσους νομίζω τα είπα. Δεν είναι τη δική μα αρμοδιότητας θέμα να το λύσουμε. Η σχέση με την πρωτοβουλία Belts and Roads. Πάλι σχετίζεται με το screening από το FDI. Δεν είναι μέσα στην ε, μελέτη. Η πρωτοβουλία αυτή, η Belt and Road, περιλαμβάνει ένα μνημόνιο κατανόησης που έχει υπογράψει η Κίνα και κάποια κράτη-μέλη. Και προϋποθέτει συνεργασία. Το screening, το πλαίσιο screening για το FDI μιλά για εξαγορές. Οπότε, σήμερα γίνεται πολλή συζήτηση για τα δίκτυα πέμπτης γενιάς, για το αν το screening του FDI θα μπορέσει να καλύψει και αυτά. Το screening μπορεί να, όπως οποιοδήποτε screening που γίνεται σε οποιαδήποτε χώρα, οποιοδήποτε screening ασφάλειας για τις επενδύσεις, μελετά τους ξένους επενδυτές που αγοράζουν μια εταιρεία ή που δημιουργούν μια εταιρεία. Δεν ελέγχει την δημόσια προμήθεια και την αγορά προμηθειών. Δεν ελέγχει τον πάροχο και το δίκτυο παρόχων των ευρωπαϊκών εταίρων, αυτό ξεπερνά λιγάκι τη δυνατότητα του screening. Αυτό που μπορεί να κάνει το screening είναι να δει του κινδύνου που μπορεί να προκύπτουν από την εξαγορά μια εταιρεία από έναν ξένο επενδυτή, ε, μια ευρωπαϊκή εταιρεία ή από τη δημιουργία μια εταιρεία δική του. Αυτό πρέπει να δούμε λοιπόν, ανεξάρτητα από το τι συνεργασία έχουμε με την Κίνα, τη Ρωσία ή οποιοδήποτε άλλο μέλο. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει κινέζικο, κινέζικη εταιρεία ή ρωσική ή η αμερικανική που αγοράζει μια ευρωπαϊκή, πρέπει να μελετήσουμε την περίπτωση αυτή, να δούμε αν υπάρχουν απειλέ, ευάλωτα σημεία, τροτά και μετά εκδίδουμε την γνωμοδότησή μα. Αυτό κάνουμε. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα συμβατότητα δηλαδή τόσο πολύ με το είναι πρωτοβουλία Belt and Road, αλλά πρέπει να δούμε κάθε μεμονωμένη συναλλαγή που γίνεται, κάθε μεμονωμένη εξαγορά για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει απειλή, δεν υπάρχει κίνδυνος. Γιατί πολλές εταιρείε είναι σε συνεργασία με την Κίνα, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη επικίνδυνες. Τις βλέπουμε ανά περίπτωση. Και γι' αυτό που είπε ο Πρόεδρος, η συμπεριφορά των ξένων άμεσων επενδύσεων σε σχέση με την επιρροή στο εργατικό δυναμικό. Δεν ήταν στο πεδίο εφαρμογή αυτό, στο φάσμα του, της μελέτης. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι η προσωπική μου άποψη. Επειδή έχω πολλά χρόνια που ασχολούμαι με τις, ε, άμεσες, με τις ξένες επενδύσεις, όχι τόσο στην Ευρώπη, σε αναπτυσσόμενες χώρες κυρίως, συνολικά ξέρουμε όλοι ότι και σύμφωνα με τα στατιστικά, οι, άμεσες, οι ξένες επενδύσεις, οι ευρωπαϊκές ας πούμε στο εξωτερικό, συνήθως συμπεριφέρονται καλά, τήρουν τους κανόνες ε, του εργατικού δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι και πιο αποτελεσματικές και προσφέρουν καινοτομία στην οικονομία, συνδέονται καλύτερα με την τοπική οικονομία. Αυτό γίνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρη εικόνα απόλυτα. Αυτό που ξέρουμε όμως σίγουρα και ίσως να είναι και το αποτέλεσμα ότι συνήθως είναι μεγαλύτερες αυτές οι εταιρείε. Ε, οι μισθοί που καταβάλλονται είναι πιο υψηλοί, αλλά τώρα για την ε, συμμόρφωση με το εργατικό, με δίκαιο της ε, χώρα χώρας, ε, εκεί δεν ξέρω να σας πω πολλά. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Κλείνουμε και το σημείο 14. Το 15 είναι το αγαπημένο μου. Είναι τα διάφορα. Δεν έχουμε όμως διάφορα. Και το 16 είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης ίντα, γιατί είναι και η τελευταία αυτή τη ε, θητείας και πρέπει να τα εγκρίνουμε τώρα. Αντιρρήσεις υπάρχουν? Όχι. Άρα εγκρίνονται τα πρακτικά των δύο αυτών ημερών και αυτό είναι και το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για την σημερινή μας συνεδρίαση και για την θητεία. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ τη γραμματεία για όλη τη βοήθεια που μας έδωσε αυτή την θητεία. So, done